και ο κύριος Κοτσολίνος συμφωνεί με αυτό, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Θα πρέπει ίσως να οργανωθούμε έτσι ώστε στην επόμενη συνάντηση να μας παρουσιάσει μια νέα έκθεση ουσιαστικά η οποία να λαμβάνει υπόψη την τελική ε, θα έλεγα επιθυμία, τις τελικές επιθυμίες των μελών της Επιτροπής. Λοιπόν, δεν θα υπάρχει ψηφοφορία για τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και περνάμε στο 9 στην απαλλαγή για το 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον Αντιπρόεδρο κύριο Στάες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. στο σχέδιο της έκθεσης που συνέταξα νομίζω ότι δούλεψα πάνω σε ένα πολύ ευρύ θέμα. Ε, κατά κάποιο τρόπο είχε χαρακτηρά αυτοκριτικής ε, η δουλειά μου αυτή ε, μια που χθες στις λεπτομέρειες του θέματος συζητήσαμε με τρεις επίτροπους το τι θα γίνει με την απαλλαγή προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η απαλλαγή είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και επομένω θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ανάλογα. Πρόκειται δε για μια προσέγγιση που και εγώ την υιοθέτησα στην εκθεσή μου. Πάντως είναι και κάπως ιδιόρυθμη αυτή η δουλειά, μια που το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει την απαλλαγή και ξεκινώ με τα καλά μαντάτα. Να τη δώσουμε την απαλλαγή έτσι προς τον πρόεδρό μας. Όμως, σε αυτή μου την έκθεση μέσα σε 30-32 σελίδες, να με τη μετάφραση, κάνω μια αρκετά επικριτική ανάλυση σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν. Και αυτά δεν τα κάνω ελαφρά την καρδία. Στηρίζομαι σε έγγραφα. Σε έγγραφα τα οποία μπορεί κανείς να τα βρει και να τα διαβάσει ή στο website της ε, Επιτροπής μας. Έχω ξανακάνει αυτή τη δουλειά, δηλαδή να κάνω έκθεση για την απαλλαγή. Αυτή τη φορά όμως η προσέγγιση είναι λίγο διαφορετική. Οπότε, θα πρέπει να βάλουμε πράγματα στι θέσει του, θα πρέπει να εξηγήσουμε ακριβώ ε, πώ έχουν τα πράγματα, τι θα πει η απαλλαγή. Διότι μπορείτε να διαπιστώσετε ότι όσον αφορά αυτή την έκθεση, έχω διατυπώσει κάποιε ανησυχίε μου, κάποιε αμφιβολίε, κάποια ερωτήματα. Οπότε και θέλω να πω πώ θα πρέπει να φροντίσουμε. Κατά πόσον. Αν Θέλουμε εξωπρεπώ να κατέβουμε στην επόμενη προεκλογική καμπάνια και να εκλεγούμε. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε κάποιους σκόπελους. Υπάρχουν κάποια θέματα δυσάρεστα, κάποια πράγματα τα οποία δύσκολα κανεί μπορεί να τα υποστηρίξει όταν κουβεντιάζει με τον κόσμο. Γιατί οι εκλογέ μα είναι και φορολογούμενοι και δηλαδή το κοινοβούλιο λειτουργεί με τα δικά του λεφτά. 1,4 δις ευρώ είναι ο προϋπολογισμός μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω, και θα μπορούσαμε να γεμίσω την αίθουσα με ψηλά τα οποία να αντιπροσωπεύουν αυτό το ποσό. Εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι το ποσό δεν είναι πενταροδεκάρε. Στη δε έκθεσή μου έχω προσπαθήσει να βάλω μια τάξη στα πράγματα. Έχω τι οκτώ πρώτε παραγράφους οι οποίε αφορούν το σύστημα διαχείρισης στο Κοινοβούλιο, την διακυβέρνηση, την εταιρική Κατόπιν έχω κάποιες προτάσεις που αφορούν την νοοτροπία που διέπει του Κοινοβουλίου, τη διαχείριση των Προέδρων, το Προεδρείο, τη Γενική Γραμματεία, του, τις Γενικές Διευθύνσεις. Και θεωρώ ότι η αφετηρία είναι μία τέτοια οτροπία η οποία διέπτει η λειτουργία μας. Έχουμε μένω σε αυτήν την εταιρική διακυβέρνηση, corporate governance στα αγγλικά. Για, και λέω για κάποιες συστάσεις που θεωρώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά το πώς θα πρέπει να γίνεται ο έλεγχος που θα πρέπει να αναβαθμιστεί η ισχύουσα διαδικασία, ε, κάτι το οποίο θέσπισε το 2002. Επομένω, ήρθε η ώρα, θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή, μια ενημέρωση. Αυτά λοιπόν ε, προτείνω. Κατόπιν έχω 12-13 παραγράφους όσον αφορά τη διαδικασία της απαλλαγής. Πρόκειται επομένω ουσιαστικά για κείμενο αυτοκριτικής επικρίνω την οικονομική μας διαχείριση. Σετάζω τις ευθύνες του Κοινοβουλίου που θεωρώ ότι είναι υπόλογο έναντι των φορολογούμενων συμπολιτών μας. Έχω δε τις παραγράφους 21 έως 24. Εκεί έχουμε την παράδοση των λογαριασμών του Κοινοβουλίου Μιλάμε για 1,4 δις ευρώ για τον προϋπολογισμό. 1% δηλαδή του προϋπολογισμού της Ένωσης. ...20% των συνολικών διοικητικών δαπανών. Επίσης, έχω κάποιες αυτοκριτικές παρατηρήσεις όσον αφορά κάποιους ε, διαγωνισμούς, τις δημόσιες συμβάσεις έχω κάνει και σε αυτό το θέμα μία σχετική έκθεση. Έχουμε κάποιες προτάσεις του κ. Κάλβεν και τις λαμβάνω υπόψη. πιστώνουμε δε ότι οφείλουμε να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα. Τι γίνεται με αυτές τις δημόσιες συμβάσεις που πρόκειται για έναν τομέα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι κάτι που άπτεται και του δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα. Πολλέ φορέ διακυβεύονται και πάρα πολύ σημαντικά ποσά. Εάν επομένω δεν είναι πολύ καλά περιχαρακωμένο, τότε ο κίνδυνο είναι να μην έχουμε εύρυθμη λειτουργία. Έχω εδώ πέρα επομένω κάποιε προτάσει προ τον Γενικό Γραμματέα. του οποίου φυσικά έχει ενισχυθεί ο ρόλος όσον αφορά τα θέματα αυτά, διότι σας ξαναλέω, οι παρατηρήσεις μου δεν ε, είναι βέλη κατά συγκεκριμένου προσώπου. Όλα αυτά τα λέω για να βοηθήσω ε, την διοίκηση και κυρίως το υψηλά στόμα της διοίκησης του Κοινοβουλίου, ούτως ώστε αυτοί οι αρμόδιοι να μπορούν να εργαστούν όπως πρέπει. Και έτσι σχολιάζω και το των δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντα όλα αυτά υπόψη ούτω ώστε να ολοκληρώσω αυτέ τι παραγράφου. Λέω λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει έλλειψη ισορροπία σε σχέση με τη συνήθη διαδικασία και από την άλλη μεριά τη διαδικασία ε, την ε, εξαιρετική, την ε, καταξιές διαδικασία κάποιων διαπραγματεύσεων και έχουμε εδώ πέρα και το θέμα κάποιου προγράμματος δράσης που θα πρέπει να προωθηθεί κάτω πάμε στους παραγράφους 49 με 59. Η διαχείριση των κινδύνων πρόκειται για κάτι που και αυτό έχει συζητηθεί με τον Γενικό Γραμματέα. Εδώ έλαβε υπόψη τόσο προβλέπει ο δημοσιονομικό κανονισμό και τι σχετικέ υποχρεώσει. Πάντοτε όμω τα πράγματα δεν είναι αγγελικά πλασμένα, διότι ε, συχνά Όλα αυτά βασίζονται σε αμοιβή εμπιστοσύνη. Έρχονται όμω οι γενικοί διευθυντέ και προβαίνουν σε κάποιες ε, δηλώσεις Και σε τέτοιες δηλώσεις οι γενικοί λένε ε, τι δεν πάει καλά στον τομέα τους. θα πρέπει κάθε Γενικός Γραμματέα πάντως να έχει κριτική και επικριτική στάση και θα πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένο για τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην υπηρεσία του. Παρακαλώ. Παράγραφο 56 έως 63. Διαχείριση κινδύνων εδώ. Είπαμε ότι θα πρέπει κάποιο πρόσωπο να οριστεί για αυτή τη δουλειά διαχειριστής κινδύνου για την ε, περίοδο 2009-2011. Αυτό το πρόσωπο θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας. Πάμε παρακάτω μετά στο 64 με 89. Είναι τη έκθεση του Ελληνικού συνεδρίου την οποία τη διάβασα με μεγάλη προσοχή. Έλαβα υπόψη τις προτάσεις του Πολιτικού Συνεδρίου. Να δω. Στην πράξη τι θα πει πολιτική ευθύνη. και συγκεκριμένα τι θα πει πολιτική ευθύνη σε περίπτωση που οι πολιτικοί λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις με οικονομικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια μέχρι 1997 έχουμε τα θέματα του ε, οικονομικού ελέγχου και ελεγκτή εσωτερικού του Κοινοβουλίου. Χαιρετίζω το ότι είναι θετικό το έργο του και στη συνέχεια, ή μάλλον μέσα σε αυτό το κείμενο ενσωματώνω, όλες τις συστάσεις επιλέξει που διατύπωσε ο οικονομικός ελεγκτής. Παρακάτω, μέχρι το 143 είναι η υπόλοιπη έκθεση και εκεί διατυπώνω τις παρατηρήσεις μου, τα συμπράσματά μου, τις επικρίσεις μου. Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία αφορούν και το Ταμείο το συνταξιδοτικό. Λέω και ότι έγινε και με την απαλλαγή λίγο πριν τις ευρωεκλογέ. Κάποια πράγματα ανεδίθησαν τότε, κάποια ζητήματα. Είπαμε για το έλλειμμα που υπάρχει στο ταμείο αυτό 28 εκατομμύρια ήταν το έλλειμμα πριν από 8 χρόνια. Όμως οι, οι επιστροφές όπως λέγονται πάντοτε δεν έγιναν όπως έπρεπε και πολλές φορές οι βουλευτές έχουν πει στην Ολομέλεια ότι αν υπάρχει πρόβλημα με το συνταξιδοτικό εκούσιο, θελούσιο, θελοντικό ταμείο, τότε υπάρχει ευθύνη που πρέπει να αποδοθεί στους διαχειριστές αλλά και σε όσους συμμετέχουν. Και θα πρέπει και εδώ την είχα την πληρώνει ο φορολογούμενος. Αυτό το λέω ξεκάθαρα στο κείμενο όπως το έχω πει και στις συναντήσεις μας. Θεωρώ διαπαράδεκτο το ότι το Προεδρείο αγνόησε την κρίση της Ολομέλειας. Σε αυτές τις επόμενες 46 τελευταίες παραγράφους υπάρχουν επικρίσεις αλλά υπάρχουν και θετικά σχόλια. Πριν από τρία χρόνια είχα μια άλλη τέτοια έκθεση όπου είχα επιμείνει στο ότι θα πρέπει να βρούμε ένα σύστημα διαχείρισης ε, φιλικό στο περιβάλλον. Οικολογική διαχείριση. Γιατί ζητάμε από βιομηχανία, γεωργία κλπ. Ζητάμε ένα σωρό πράγματα τόσο ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όμως θα πρέπει να φροντίσουμε και τα του οίκου μας. Να κάνουμε τα ίδια και στο περιβόλι μας. Ε, έχουμε αυτούς τους στόχους για το 2020, δηλαδή μείωση των εκπομπών, ε, ο στόχος του 30%. Διαπιστώνω επομένω κάποιες θετικέ εξελίξεις. Κάνουμε εξοικονόμηση στην ηλεκτρική ενέργεια. 25% σε τρία χρόνια μειώσαμε την ηλεκτρική ενέργεια. Έχουμε ανακύκλωση των ε, απορριμμάτων και 50% μειώθηκε το βουνό των σκουπιδιών. Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Λουξεμβούργο. Έχουμε ηλεκτρική ενέργεια πράσινη που χρησιμοποιούμε. Πολύ θετικά όλα αυτά τα στοιχεία. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε στους ε, συμπολίτες μας, τους φορολογούμενους. Έχουμε βέβαια και κάποια αρνητικά σημεία. Δεν χρησιμοποιούμε υβριδικά αυτοκίνητα. Ε, inzet op het, ε, op het vervoer, het individuele vervoer van... Και Έχουμε επίσης ε, ε, η κάπως υπερβολική χρήση ε, για αυτές τις λιμουζίνες που μεταφέρουν έναν έναν τους βουλευτές. Τα είχαμε πει και πέρσι. Είχε γίνει η αναθεώρηση του καθεστώτος του βουλευτή επί τη βάση του εσωτερικού ελέγχου που είχε γίνει πριν από δύο χρόνια. Τώρα Έχουμε αναθεώρηση, επίσης ενημέρωση του καθεστώτος και να δούμε εάν τώρα λειτουργεί ευρυθματό σύστημα, εάν πετυχαίνουμε τους στόχους που είχαν τεθεί. Να δούμε αν μπορούμε να συνεχίσουμε την ίδια ρότα ή αν πρέπει να επιφέρουμε και περαιτέρω βελτιώσεις. Να μην σας πω και λεπτομέρειες, μια που κάπως πιέζει ο χρόνος, αλλά για να μπορούμε να εγγυηθούμε ε, την καλύτερη των πραγμάτων θα πρέπει να λειτουργεί η δίκηση με τρόπο διάφανο και πριν γίνει η μετάφραση του κειμένου ζήτησα από κάποιους υψηλόβαθμους υπαλλήλους μας να μου πούν τις παρατηρήσεις τους. Ε, με κάποιες συμφώνησα, με άλλες δεν ε, συμφώνησα με κάποιους διαφώνησα, με κάποιους διαφώνησα ε, σε ιδεολογική βάση. Πριν από δύο εβδομάδες δε, συνδύθηκα στο Στρασβούργο με τους σκιώδεις συζητητές. Έλαβε υπόψη κάποιες παρατηρήσεις τους, ε, ας πούμε ο κύριος Γκέρ Μπράντι, είπε ότι πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί σε μερικά σημεία Έχουμε όμως κάποιες τροπολογίες θα τις συζητήσουμε Περιμένω πώς και πώς να τα συζητήσουμε τα των τροπολογιών οι οποίες 2 Μαρτίου πρόκειται να συζητηθούν στην συνάντησή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα ξεκινώντας ε, να ε, εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον κύριο Στάς για αυτά που μας είπε και να ευχαριστήσω και αυτούς οι οποίοι τον βοήθησαν στην προσπάθειά του. Είχαν ε, το θάρρος να βάλουν γραπτά κάποια πράγματα που ορισμένοι ίσως δεν θέλουν να ακούσουν, λέει ο κύριος Γκεμπραντή. Ιστορικά το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζει στον τομέα αυτό δύο βασικά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι οι αρμοδιότητές του. Τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα με τη συνθήκη της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο απέκτησε ουσιαστικές αρμοδιότητες. Δεύτερο ιστορικό πρόβλημα είναι τα ε, χρηματοπιστωτικά σκάνδαλα. Πολλά έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια βέβαια. Το θέμα του υπολόγου των πολιτικών ομάδων, η ευθύνη, εν πάση περιπτώσει, η απολογιστική των πολιτικών ομάδων. Η εσωτερική έλεγχη επίσης ε, είναι πολύ πιο ανεξάρτητη από ό,τι στο παρελθόν. Υπάρχουν πολλές επιστροφές οι οποίες γίνονται άμα την παρουσιάση δικαιολογητικών και όχι εφάπαξ πληρωμές. Γενικά τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία πρέπει να πάνε καλύτερα. Εδώ και λίγες εβδομάδες είχαμε μια συνάντηση των συντονιστών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής είπα ότι θα πρέπει να σημειώσουμε θα έλεγα με κάποιο έντονο τρόπο τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας για να βρούμε τρόπους βελτίωσης του Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με τον κύριο Στάς για την σωστή διακυβέρνηση και διαχείριση ε, του Κοινοβουλίου μας και θα μπορεί να υπάρξουν σημεία βελτίωση. Σε ένα δεύτερο σημείο είναι το θέμα της διαφάνειας. Θέλουμε πράγματι να γίνουμε καλύτερα κατανοητοί από τους εκλογείς μας. Εάν ναι, τότε θα πρέπει να είμαστε περισσότερο διαφανείς. Διαφανής σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι διαφανές 100% το χρηματοδοτικό της, το, ο, ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι εργασίες μας. Νομίζω ότι και το ύφο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σαν υπεύθυνοι της Επιτροπής ε, ε, για τον έλεγχο του προπολογισμού δεν πρέπει να δίδουμε την εντύπωση ότι όλα πάνε χάλια και ότι τα χρήματα δαπανώνται άσκοπα. Στην καλύτερη περίπτωση. Να πούμε όμως ότι παράλληλα με τις βελτιώσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει απαιτούνται συμπληρωματικές προσπάθειες. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Τέλος, μια τελευταία παρατήρηση. Υπάρχει μια αναφορά τα αυτοκίνητα. Ο κύριος Στάς προτείνει στο να περάσουμε σε υβριδικού τύπου αυτοκίνητα. Δεν είναι κακή ιδέα βέβαια. Σαν Ολλανδός θα έλεγα ότι καλό θα είναι να θέσουμε στη διάθεση των βουλευτών ποδήλατα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω πολύ πιο εύκολα τα ποδήλατα στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες και θα καταθέσω τροπολογία για την χρήση ποδηλάτων. κύριος Ήταλα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τον εισηγητή η συνεργασία που πρόσφερε ήταν θετική και ανοιχτή. Συμφωνώ και με την προσέγγιση του θέματος που επέλεξε από την σκοπιά δηλαδή των φορολογουμένων αφού μιλούμε εν τέλει για χρήματα των φορολογουμένων δεν δικά μας αυτά τα χρήματα που θα πανούμε και έτσι πρέπει να το δούμε εγώ θα ήθελα να υπάρχει ακόμα περισσότερη διαφάνεια μένουν ακόμα πολλά πράγματα να γίνουν για παράδειγμα, οι διαδικασίε για τη λήψη των αποφάσεων. Προπολογισμό του 2008. Ιδιαίτερα περίπλοκη διαδικασία. Η Επιτροπή Προπολογισμών αποφασίζει το Α, το Προεδρείο αποφασίζει το Β. Και δεν είναι πλέον πολύ ξεκάθαρο ποια απόφαση έχει προτεραιότητα. Υπερτερή. Τώρα, επί της εκθέσεως του κυρίου ε, Στάς. Εγώ νομίζω ότι ορισμένα τμήματα πρέπει να διαγραφούν. Υπάρχουν και ορισμένες ερωτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλίου. Κυρίως ό,τι αφορά την πολιτική ακινήτων. Πληρώνουμε υπερβολικά πολλά για τα ακίνητα. Για το κτίριο του Στρασβούργου. Το αγοράσαμε, λειτουργεί, αλλά δεν λειτουργεί καλά χρειάστηκε να αφαιρεθεί ο αμίαντος. Αυτά έγιναν εν μέρη και με συμμετοχή του Κοινοβουλίου, άρα με χρήματα των φορολογουμένων, ενώ θα έπρεπε να τα είχε κάνει ο Δήμος Στρασβούργου. Το άλλο είναι το κέντρο επισκεπτών. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ, να έχει τελειώσει πολύ νωρίτερα. Υπάρχουν καθυστερήσει και εδώ κάποιο πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε. Θεωρώ ότι δαπανώνται, ότι σπαταλώνται χρήματα των φορολογουμένων πρέπει να απαντήσει πιο ξεκάθαρα ο Γενικός Γραμματέας. Δυνατότητες βελτιώσεων. Βελτιώσει έχουν υπάρξει. Αφού τώρα γίνεται απόδοση λογαριασμών στη βάση των πραγματικών δαπανών. Αλλά για τους επισκέπτες όχι. Εκεί μπορεί να βελτιωθούν κάποια πράγματα. Τώρα για το κανάλι τηλεόρασης του Κοινοβουλίου αποδίδει η επένδυσή μας. Πόσους θεατές διαθέτει το κανάλι αυτό. Πώς μπορεί να προσελκύσει περισσότερους τηλεθεατές το κανάλι αυτό. Εξάλλου, συμφωνώ με τον εισηγητή όταν θέτει το ερώτημα τι γίνεται με την φήμη του Κοινοβουλίου. Μιλούμε εδώ για χρήματα αλλά προς τα έξω δεν καθίσταται σαφές ότι τώρα είναι καλύτερη η κατάσταση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα χρήματα που κακώς δαπανήθηκαν πρέπει να τα ανακτήσουμε. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να τα ανακτήσουμε. Πρέπει να τακτοποιήσουμε τα του οίκου μας πρώτα. Ακόμα και αν είναι μικρά σχετικά ποσά, Πρέπει κάτι να γίνει για να ανακτηθούν. Ένα τελευταίο. Συμφωνώ με τον εισηγητή που λέει ότι πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Όταν ζητούμε από τους πολίτες να κάνουν αλλαγές ε, στη ζωή τους, να τις κάνουμε τις αλλαγές αυτές και εμείς. Η υβριδικά αυτοκίνητα για παράδειγμα. Βέβαια, κοιτάξτε, άμα βρέχει καταροκτόδοξα έξω δεν θα πάρω το ποδήλατο. Αλλά υπάρχουν και τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας. Στην Φιλανδία, στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε και εισιτήρια του μετρό. Και από τότε που έγινε αυτό, οι βουλευτές χρησιμοποιούν όλο και λιγότερο τα προσωπικά τους αυτοκίνητα. Η κυρία Κρέσλε. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Μπάρτ, πραγματικά σκοτώθηκε στη δουλειά. Δεν θυμάμαι να έχω διαβάσει άλλη φορά τόσο μακροσκελή έκθεση. Ίσως όμως και να μην θυμάμαι τόσο καλά. Εγώ βέβαια δεν είμαι από τα πρόσωπα εκείνα που αποφεύγουν τους καυγάδες. Ορισμένου καυγάδε θα προτιμούσα ωστόσο να του αποφύγω, για παράδειγμα με το Προεδρείο του Κοινοβουλίου, σχετικά με το ποιο είναι αρμόδιο να λάβει ποιε αποφάσει και ποιο έχει υποχρέωση να αναλάβει ποιε ευθύνε. Την έχουμε διεξαγάγει την συζήτηση αυτή παλαιότερα κατά επανάληψη. Αλλά εδώ δεν την περιλαμβάνει. Αποφασίζει λίγο αυθαίρετα, θα έλεγα, ποιο πρέπει να αποφασίζει τι. Με λυπεί λίγο αυτό, διότι η συζήτηση αυτή έχει γίνει στο παρελθόν. Και υπάρχουν ορισμένα μεγάλα θέματα όπως 2007-2008. Τα μεγάλα θέματα συγκρούσεων δεν περιλαμβάνονται στην έκθεση. Η έκθεση αυτή που έχει και κάπως θεωρητικό χαρακτήρα. Όταν μιλώ για τέτοια θέματα συγκρούσεων εννοώ για παράδειγμα το αθλητικό κέντρο όπου εκεί μαλώσαμε πολύ με το Προεδρείο και τελικώς ιτήθη το Προεδρείο. Επίσης, το staff screening που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα μέσα που χρησιμοποίησε και εμείς ωστόσο αρνούμαστε να υιοθετήσουμε τα ίδια μέσα και να κάνουμε το ίδιο screening. Θα ήθελα να το δω αυτό στην έκθεσή σου. Ένα άλλο που δεν με ναι, βρίσκει σύμφωνη είναι ένα είδο γενικής υποψίας που πλανάται πάνω από τα κεφάλια όλων σχετικά με το πώς διαχειριζόμαστε τα χρήματα. Αυτή η γενική υποψία δεν είναι σωστή. Η αναθεώρηση του γραμματιακού επιδόματος είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που επέτυχε η ε, παρούσα Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού. Τώρα να έρχεσαι και να λες ότι δεν, πρέπει να υπάρξει καμία αύξηση, αυτό δεν με βρίσκει σύμφωνη. Εγώ χρειάζομαι αύξηση του γραμματιακού επιδόματο διότι χρειάζομαι περισσότερους συνεργάτες για να μπορώ να εργάζομαι σωστά. Για την ώρα έχω εξαντλήσει κάθε όριο του γραμματιακού επιδόματό μου. Αυτό λοιπόν που λες εδώ δεν μου αρέσει. Τώρα ένα άλλο. Λες ότι είμαι αποδέκτης επιδοτήσεων ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ έχω την αποζημίωσή μου και αποζημίωση από τη γερμανική Bundestag, γιατί έχω παραμείνει στο παλαιό σύστημα. Γιατί λοιπόν λες εδώ ότι είμαι τελικός αποδέκτης επιδοτήσεων. Αν εννοείς το γραμματιακό επίδομα, αν πρέπει να δημοσιεύσω αυτά στο διαδίκτυο μαζί και με τα έξοδα ταξιδιού τους όπως ζητούν ορισμένοι δημοσιογράφοι. Εγώ βρίσκω ότι είναι υπερβολικά τολμηρές αυτές οι διατυπώσεις διότι αν εγώ ως Ευρωβουλευτής είμαι τελικός αποδέκτης επιδοτήσεων τότε όλοι οι ευρωϊπάλληλοι είναι τελικοί αποδέκτες επιδοτήσεων και χαίρομαι ήδη από τώρα διότι θα πρέπει όλοι να δημοσιεύσουν τις απολαβές τους στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε λίγο για την σύνταξη. Το άλλο είναι αυτή η εκδρομή για το σκι. 84.000 ευρώ είναι απίστευτα. Τα μικρά ποσά είναι αυτά που είναι επικίνδυνα. Και εδώ πρέπει να τοποθετηθούμε. Εμεί θα καταθέσουμε τροπολογία λοιπόν και θα ζητήσω ήδη από του συναδέλφου να την υποστηρίξουν. Τα κλασικά θέματα, τα κλασικά δημοσιονομικά θέματα λοιπόν, βρίσκουν να λείπουν κάπως από την έκθεση και θα τα συμπληρώσουμε εμεί. Η κυρία Ερτσόκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον κύριο Στάσο, κύριο συγγήτρια των Σοσιαλιστών, καθώ και του άλλου κυρίω συγγητέ για την καλή συνεργασία, για προ την κατεύθυνση να επιτύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, μια καλή έκθεση για την απαλλαγή αυτή. Εμεί οι Σοσιαλιστέ χαιρόμαστε για την πρωτοβουλία του κύριου Στά να μην παραμείνει μονάχα στην απαλλαγή, αλλά να κάνει ένα είδος ε, πενταετούς σχεδίου για το που θέλει να φτάσει το Κοινοβούλιο σε πέντε χρόνια στη διάρκεια της παρούσας θητείας δηλαδή. Και νομίζω ότι πράγματι η παρούσα διαδικασία απαλλαγή είναι και σωστός τόπος για να διατυπωθούν ορισμένοι στόχοι για τα επόμενα πέντε χρόνια. Και με ικανοποιεί αυτό και ιδίω όταν οι στόχοι αυτοί έχουν το νόημα περισσότερης διαφάνειας, περισσότερης αποτελεσματικότητας και τελικά περισσότερων επιτυχιών για όλου μας. Χαιρόμαστε λοιπόν για την έκθεση. Υπάρχουν ορισμένα θέματα που θα συζητήσουμε και οι ανθρώπινοι και οι δημοσιονομικοί και οι φυσικοί πόροι του Κοινοβουλίου πρέπει να εκτιμώνται, να αξιολογούνται ισορροπημένα για το μέλλον και ο εσωτερικός έλεγχος του Κοινοβουλίου πρέπει να ενισχυθεί γιατί είναι το πιο οριζόντιο εργαλείο, ο πιο, ο πιο οριζόντιος μηχανισμός εκεί μπορούν να συνεργαστούν όλες οι γενικές διευθύνσεις του Ευρωκοινοβουλίου και να στοχευτεί καλύτερα η αξιολόγηση του κινδύνου. Νομίζω ότι αυτό θα με ενδιέφερε περισσότερο. Συμφωνώ με τους κυρίους Ιταλά και Κρέσλε ότι η πολιτική κινήτων πρέπει να γίνει με καλύτερο τρόπο. Ας το πούμε έτσι. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό. Και το αθλητικό κέντρο βέβαια αποτελεί τμήμα της πολιτικής ακινήτων. Υπάρχει ένας αριθμός θεμάτων της έκθεσης που αναφέρεται στις πολιτικές ομάδες. Εγώ πρότεινα να πάμε να βρούμε τους ταμείες και ενδεχομένω τους γενικούς γραμματείς των πολιτικών ομάδων, το δέχτηκαν αυτό και οι οι να μας δώσουν μια ιδέα πού βρίσκουν ότι μπορεί να γίνει κάποια βελτίωση. Και μπορούν τότε να διατυπωθούν με καλύτερο τρόπο οι παράγραφοι αυτές. Αλλά πάντως χαιρόμαστε που θέτεται τα θέματα αυτά. Θέλουμε να ενισχυθεί η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Βλέπουμε ωστόσο ταυτόχρονα ότι δεν μπορεί να είναι η αστυνομία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροπία μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και του εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να κάνει τον πραγματικό έλεγχο. Εμείς θα διατυπώσουμε τροπολογίες για να βελτιωθεί έτσι περαιτέρω η έκθεση. Ευχαριστώ και το ελεγκτικό συνέδριο διότι η δική τους έκθεση μας βοήθησε πολύ. Γενικά νομίζω πρέπει να διατηρήσουμε ένα θετικό πνεύμα, διότι επιτεύχθηκαν σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, για τους κοινοβουλευτικούς συνεργάτες. Ας μην το υποτιμούμε αυτό. Και βέβαια, όταν έχουμε την ευκαιρία να λέμε στο κοινό ότι στην τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο το Κοινοβούλιο κινήθηκε προ τι σωστέ κατευθύνσεις. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Να λέμε δηλαδή και τα καλά νέα στον κόσμο, όχι μόνο τα άσχημα. Σας ευχαριστώ και αρκούμε σε αυτά. Η κυρία Ματιού. Ε, και εγώ, όπω και όλοι συναδελφοί, να συγχαρώ τον εισηγητή, διότι ήταν εξαιρετική η έκθεσή του Και θέλω να σταθώ σε δύο σημεία της έκθεσης. Με ενδιαφέρει πρώτα πρώτα το τι γίνεται με τις ομάδες των επισκεπτών που προσκαλούμε στο Κοινοβούλιο. Δικαιούμεθα δύο ετησίως σύμφωνα με το ισχύον σύστημα το οποίο όμως δεν εξυπηρετεί τόσο πολύ την προβολή μας. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι επισκέπτες οι επικεφαλής τους αμείβονται σε μετρητά από το κοινοβούλιο αυτό δεν, δεν βοηθάει την προβολή μας γιατί είναι κάτι λέμε το οποίο μας ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ όλοι οι συναδέλφοι. Εγώ όμως οφείλω να σας πω ότι για κάθε ομάδα επισκεπτών που έρχεται ε, θα πρέπει να αυτό το πρόβλημα, ότι δηλαδή η εντύπωση είναι πάρα πολύ αρνητική σε σχέση με αυτά τα χρήματα τα οποία πληρώνονται σε μετρητά. Τα μισά πάνε τόσο με έμβασμα και τα άλλα μισά στον επικεφαλής της ομάδας σε μετρητά. Αυτό είναι πάρα πολύ αρνητικό για την εικόνα του Κοινοβουλίου. Εγώ πάντα τους καλώ στο Στρασβούργο, πάμε στα Βόσγια και κάθε φορά 35 ευρώ περίπου να πληρώσω για τα γεύματα και λέει ο κόσμος «Ε, τι θα γίνει με κάποια διαφορά πολλές φορές προκύπτει όταν κάποιος μένει κοντά στο ασβουργείο γιατί πολλές φορές βγαίνει ανά ομάδα επισκεπτών ένα, ένα ποσό 800.000 ε, ευρώ που θα πρέπει να καταβληθούν για, για τη μεταφορά ε, οπότε υπάρχει ένα μικρό ποσό το οποίο λείπει, θα πρέπει να συμβάλλει ο κόσμος, αλλά αυτό φέρνει μεγάλη δυσαρέσκεια. Και βεβαίω και είναι υποχρεωσή μας να καλούμε τον κόσμο, αλλά είδατε, βγαίνει δυσαρέσκεια από αυτή την κατάσταση. Άρα, τελικά, ε, δεν βγαίνουμε κερδισμένοι από αυτή την υπόθεση, επομένως, ας τους ε, αποζημιώνουμε επί τη βάση κάποιες απόδειξες και έτσι θα είναι το ακριβές ποσό ας πούμε για τα γεύματα, για τη μεταφορά και όταν υπάρχει κάποιο υπόλοιπο πού να επιστραφεί αυτό ασχολούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι πάνε να ε, να ασχοληθούν με αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές που, που μένουν πιο κοντά, άλλοι μένουν πιο μακριά και έτσι αυτό εξορροπείται κάπως. Αλλά όμως παραμένει πρόβλημα. Τι λες να κάνω, θες εσύ να το, το βάλεις αυτό το θέμα μέσα στο κείμενό σου, να κατεβάσω κάποιες τροπολογίες. Γιατί είναι αποτελεί πρόβλημα. Μπορεί αυτά να είναι λεπτομεριακά θέματα, αλλά ε, είναι πάρα πολύ αρνητικό το, να φεύγουν κρατώντα ένα μάτσο χαρτονομίσματα, να φεύγουν το κοινοβούλιο. Πολύ κακό για την εικόνα μα, πρόεδρο. Eh, Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κύριο Ντόιτς και εγώ να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Στάς και να σταθώ σε πέντε παρατηρήσεις. Πρώτα πρώτα. Μιλούμε για την διαφάνεια σε σχέση με τη διαδικασία ζώη της απαλλαγής. Και θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση. Az Európai Unió 27 tagországában 27 Συνεχίζει ο μιλητής. Μιλούμε για 27 χώρες μέλη. Έχουμε επομένως 27 εθνικά κοινοβούλια. Να κάτσουμε επομένως και να δούμε Τι γίνεται με την διαφάνεια στα ελληνικά κοινοβούλια. Να κάτσουμε και να βρούμε πού υπάρχει περισσότερη διαφάνεια, δηλαδή η αρίστη πρακτική. Κατόπιν αυτή τη σύγκριση, λοιπόν, εντοπίζουμε ποιος είναι ο καλύτερος και προσπαθούμε να υιοθετήσουμε αυτό τα οποία κάνει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν λέω τώρα για να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, λέω απλώς ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει πιο καλά το Κοινοβούλιο ή η Ένωση. Αρκεί επομένως να υιοθετήσουμε μια πετυχημένη συνταγή που ε, την έχει κάποιος άλλος κάπου αλλού. σε άλλα σημεία τώρα. Να σας πω και εγώ για τα θέματα που με ενδιαφέρουν, όπως έχουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Ανέκαθεν, με ενδιαφέρουν τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ας πούμε το να μην τυπώνουμε χωρίς να χρειάζεται πολλά έγγραφα από το ίντερνετ, από το email, γιατί πολλές φορές γεμίζουμε με τέτοια άχρηστα ε, print-out. Ε, έτσι καλώ ξέρετε, δαπανούμε τόσα χρήματα ούτως ώστε να βελτιώνουμε την πληροφορική στην Ένωση και στο Κοινοβούλιο. Αλλά ταυτόχρονα να κάτσουμε και να έχουμε υπόψη πόσο χαρτί τυπώνεται για μία συνεδρίαση, Φερρυπίν. Μιλάμε για ποσότητες πολύ μεγάλες. Α πούμε, χωρί να χρειάζεται τυπών αντέγραφα για του βουλευτέ οι οποίοι αδυνατούν να προσέλθουν στη συνεδρίαση. Είναι σημαντικό αυτό για το περιβάλλον. Και. Επομένω, να κάτσουμε να δούμε πόσα κιλά χαρτιού τυπωμένου αντιστοιχούν ανά βουλευτή. χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων, ειδικών συμβούλων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό δεν είναι κακό. Όμως, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα website όπου κανείς θα μπορεί να βρει τις μελέτες, τις γνώμες, τις γνωμοδοτήσεις αυτών των ειδικών, των εμπειρογνωμόνων. Έτσι ίσως προκύψει κάποια οικονομία γιατί έτσι θα αποφύγουμε να έχουμε για το ίδιο θέμα περισσότερες μελέτες και ανάθεση αυτών σε περισσότερους εμπειρογνώμονες. Για την κυρία Γκρέσλε θέλω να πω ότι βεβαίως μας απασχολούν και τα νέα θέματα και τα παραδοσιακά και γι' αυτό και έλαβε υπόψη δεν θέλω να ξαναπούμε τα ίδια. Όμως υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί στο κείμενο της έκθεσης. Να κάτσουμε για να δούμε ειδικότερα κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις επιτροπές. Στις επιτροπές αποφασίζουν κάποιοι οι οποίοι έχουν προέλθει από κάποιες άμεσες εκλογές. Όμως στις επιτροπές τις κοινοβουλευτικές αποφασίζουν και κάποιοι υπάλληλοι. Το σύστημα λειτουργεί καλά όταν είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες εκάστου. Οπότε και μπορούμε εμείς να ξέρουμε ποιες είναι οι αποφάσεις που παίρνουν οι αιρετοί, οι βουλευτές δηλαδή, και ποιες είναι οι αποφάσεις που πρέπει και δίνονται να λαμβάνουν οι υπάλληλοι. Νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά ξεκαθαρισμένα και αυτό θα, θα πρέπει να κάνουμε. Όταν ε, κάνουμε την απαλλαγή, τη διαδικασία της απαλλαγής, για διάφορους ε, οργανισμούς και θεσμικά όργανα. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κάποια έγγραφα, κάποιες γνωμοδοτήσεις και θεωρούμε ότι οι συστάσεις έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικό. Όταν λοιπόν καταρτίζουμε κάποια έκθεση για τη διαφάνεια, για τον προϋπολογισμό, ε, για τη σύνομη λειτουργία κάποιου οργανισμού, Πάρα πολύ καλό είναι αυτό το οποίο κάνουμε. Όμως θα πρέπει όλα όσα συστήνουμε στους άλλους θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε και στο περιβόλι μας και στο σπίτι μας. Να δούμε τι πρακτική ακολουθείται στη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Μήπως εμείς κάνουμε κάτι που έχουμε επικρίνει σε κάποιο άλλο θεσμικό όργανο. Να μην είμαστε δηλαδή πιο αυστηροί με τους άλλους παρά με τον εαυτό μας. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή, αλλά να του ζητήσω και συγγνώμη γιατί ήρθα με κάποια καθυστέρηση και έχασα ένα μέρος της ομιλίας του γιατί ήμουν σε άλλη συνεδρίαση. Αλλά αυτό που θέλω να πω τώρα είναι ότι κυρίως με ενδιαφέρουν τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά ιδρύματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο τρόπο με τον οποίο γίνεται η χρηματοδότηση αυτή δεν είναι πολύ διαφανής. Παράδειγμα, για το 2008 που είναι το έτος που μας ενδιαφέρει, το Προεδρείο απεφάσισε κάποια στιγμή να διαθέσει 6 εκατομμύρια ευρώ επί για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα χωρίς να προσθέσει κάποια αιτιολόγηση. Είπε, ο ναι, έρχονται οι ευρωεκλογέ και πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον του κοινού για προσέλευση στις ευρωεκλογέ. Χωρίς άλλη εξήγηση. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει παρά μόνο ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, τα οποία βέβαια διευθύνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, χρειάζονταν περισσότερα χρήματα. Και μιλούμε για μεγάλα ποσά μεταξύ του 2004 και του 2008. Μόνο για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα μιλούμε για 60 εκατομμύρια ευρώ. 18 εκατομμύρια ευρώ το 2010 για κόμματα και ιδρύματα. Δύο ερωτήσεις και δύο προτάσεις. Πρώτο, ελείπει πας έλεγχος για την δαπάνηση αυτών των μεγάλων ποσών που καταλήγουν στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και στα πολιτικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει έλεγχος. Για την ώρα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Παράδειγμα, έθεσα ορισμένες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με την χρήση των κονδυλίων για το 2008. Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα οφείλουν να υποβάλουν στο Κοινοβούλιο ετησίως έκθεση ελέγχου μέσα στο εξάμεινο που ακολουθεί το τέλος του έτους. Διατύπωσα για το Πράσινο Ίδρυμα ότι δεν υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση. Άρα δεν έγινε και έλεγχος από πλευράς Κοινοβουλίου. Ουδής το διεπίστωσε αυτό μέχρι ό,τι εγώ κατέθεσα σχετική κοινοβουλευτική ερώτηση. Αυτό δείχνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει σημαντικές πληρωμές, σημαντικές καταβολές από χρήματα των φορολογουμένων, προβλέπει υποτίθεται κάποιους ελέγχους, στην πραγματικότητα αυτοί οι έλεγχοι δεν πραγματοποιούνται. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο εισηγητής και βέβαια η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού θα πρέπει να εξετάσουν το νόημα ή και την έλλειψη νοήματος των ποσών αυτών που γίνονται όλο και μεγαλύτερα και που κατευθύνονται στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων, κομματικών ιδρυμάτων. Από το 2004 έχουν αυξηθεί εκθετικά τα ποσά αυτά. Και εγώ δεν βρίσκω να υπάρχει καμία απολύτως αιτιολόγηση. Ευχαριστώ. Ως νέο μέλος της ε, Επιτροπής θα ήθελα να αντισταθώ στον πειρασμό να υπησέλθω σε λεπτομέρειες. και να επεκταθώ σε αυτά. Γι' αυτό θα περιοριστώ σε δύο θέματα. Διάβασα στην εκθεσή σας ότι ακόμα δεν έχει λήξει το θέμα του αμοιάντου στους διαφόρους χώρους του Κοινοβουλίου ότι ναι μεν προσωρινά έχει διευθετηθεί αλλά βλέπω εδώ μία φράση ότι ναι μεν έχει περικλειστεί ο αμίαντος και δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο. Αυτό σημαίνει όμως ότι μπορεί κάτι να προκύψει στο μέλλον. Χρειάζομαι περισσότερες Λεπτομέρειε, διότι θεωρώ ότι είναι ένα βαρύτατο πρόβλημα, ίσω ε, μάλιστα μαζί με άλλα προβλήματα τα οποία δεν μπορώ εγώ να αξιολογήσω τόσο καλά όπω ο προλαλή σα συναδελφό μου, αλλά το γεγονό ότι ίσω εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία των βουλευτών και των εργαζομένων στα ευρωπαϊκά όργανα. Θα ήθελα λοιπόν κάποια απάντηση εκεί. Δεύτερο, παρακολούθησα τα όσα είπε η κυρία Γκρέσλε, γιατί για μένα ήταν νέα τα στοιχεία αυτά Χαίρομαι που έφυξε το θέμα. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. σε ό,τι αφορά τους χαρακτηρισμούς που δίνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τα καθήκοντα που ασκεί, αλλά για παράδειγμα και το πώ λειτουργεί ε, πάνω σε προσωπικό και ενώ ιδιαίτερα του κοινοβουλευτικού βοηθού και το καθεστώ του. Τώρα, για τι ομάδε επισκεπτών. Δεν είναι απαραίτητο οι συνεργάτες σας να δίνουν στα χέρια των επισκεπτών χρήματα σε ρευστό. Εγώ γνωρίζω από κάθε είδους διοίκηση ότι εδώ και χρόνια μπορεί να γίνεται και πίστοση λογαριασμού. Ίσως χρειάζεται καλύτερη εκπαίδευση των συνεργατών του Κοινοβουλίου για το πώς μπορούν να γίνουν αυτό, αυτά τα πράγματα. Πραγματικά, εάν δίνονται φάκελοι με χρήματα, αυτό είναι μοιραίο λάθος. Ο κύριος Σάρμας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν επιθυμείτε να παρέμβετε... Δεν έχω παρατηρήσει. Για μα το κείμενο του κ. Στάς είναι πηγή έμπνευση. Απλώ να σα πω όσον αφορά τα τρία σημεία τη έκθεση. Α πούμε πρώτα-πρώτα τι δημόσιε συμβάσει. Το κατά πόσο είναι εξαντλητική η αιτήσια έκθεση των Γενικών Διευθυντών του Κοινοβουλίου και τις ε, δαπάνες για τα πολιτικά κόμματα. Εμείς παρακολουθούμε αυτά τα θέματα επίσης όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα. Φέτος κάναμε μια έρευνα την οποία και θα δημοσιεύσουν αφορά το 2009. Πρόεδρος. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω κλείνοντας τον Αντιπρόεδρο γιατί θεωρώ ότι επετέλεσε αξιόλογο έργο ε, με οξυδέρκεια, ε, εμβάθυνε και ε, νομίζω ότι πάρα πολύ εύστοχα δεξιά δύο πραγματικά ζητήματα να λάβουμε υπόψη το θέμα των επισκεπτών είναι θέμα διαφάνειας και επίσης τα της πολιτικής των ε, κτηρίων, των ε, ακινήτων. Γιατί μην, μην ξεχνούμε τι έγινε στο Στρασβούργο που κατέρευσε το, το κτίριο. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ένα σωρό καταγγελίες όσον αφορά τα τεράστια ποσά τα οποία δαπανούμε για τα κτίρια και σε σχέση με τα όσα δαπανούμε για την ε, μετακίνηση από Βρυξέλλες προς Στρασβούργο. Και μερικοί από κάποιε χώρε πρέπει να πάρουν τρία-τέσσερα πάνε για αυτό στο Στρασβούργο. Οπότε μπορώ να ευχαριστήσω τον κύριο Στά. Βρισκόμαστε πίσω όσον αφορά το πρόγραμμα και πάμε στο επόμενο σημείο τη μέσα διάταξη που είναι η απαλλαγή 2009 ε, για τον προπολογισμό τη Ένωση οπότε και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά συμβούλιο, οκέ, δικαστήριο. Α, να απαντήσω στις ερωτήσεις, λέει ο κύριος Στάς. Όχι, πρόεδρε. Δεν θέλω να παρελκύσω τη διαδικασία. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, αλλά υπάρχουν κάποια θέματα. Όταν μου τον ερωτήσουν. Οπότε δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τις παρατηρήσεις τους. Και με τις τροπολογίες εκεί θα είναι τα πράγματα ξεκάθαρα μια που θα είναι διατεπόμενη γράφος Ευχαριστώ την κυρία Γκρέσλε επίσης όσον αφορά τα όσα είπε. Η κυρία Χέρτσοκ μας είπε για τη συνεννόηση με τους σκιώδεις ηγητές. Φαν Χέκια για τις πολιτικές ομάδες και ιδρύματα. Θα πρέπει όντως εδώ να προβληματιστούμε, να συνοηθούμε με τους ταμείες, τους υπεύθυνους οικονομικούς των πολιτικών κομμάτων, γιατί κάποια πράγματα επιδέχονται ε, βελτίωση. Κύριε Φανχέκε, κοιτάξτε καλά τι λέω στο σημείο αυτό που θίξατε. Τι λέω στην παράγραφο 88. Όχι, 98 έως 125. Νομίζω ότι επικρίνω αρκετά τις ε, ληφθήσεις αποφάσεις όσον αφορά τα οικονομικά των ε, πολιτικών κομμάτων αλλά και ιδρυμάτων. Πολλές φορές έχει αποφασίσει το Προεδρείο επ' αυτών ε, χωρίς συζήτηση, κάτι το οποίο επιδέχεται και αυτό διόρθωση. Μίλησατε για έξι εκατομμύρια. Αυτό δεν είναι για πολιτικά κόμματα, προσοχή είναι για τι πολιτικές ομάδες. Ο δε σχετικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται όπως γίνεται και στα εθνικά πολιτικά κόμματα, γιατί ξέρετε ε, υπάρχει διαφορά σε σχέση με όσα γίνονται ε, στα κράτη-μέλη σε σχέση με όσα γίνονται στο κοινοβούλιο. Έχουμε επίση και μία έκθεση που συνδέεται για αυτό το λόγο. Οπότε και συμφωνώ με τις προτάσεις σας. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν κάποια σημεία. Επίσης μας ε, είπατε και για εκείνο το πράσινο ίδρυμα Ναι, είναι κάτι το, όπου είμαστε μπλεγμένοι και εμεί, ω πράσινοι και εγώ ήμουν ο πρώτο που επέκρινα και είπα ότι ο πρώτο πρέπει δεν είναι το καλό παράδειγμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με την πολιτική των κτηρίων. Εγώ είμαι υπεύθυνη για το θέμα αυτό και θα ασχοληθώ νομίζω και στο άμεσο μέλλον με την υπόθεση αυτή και με το Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούμε να συμφωνήσουμε σε έναν κατάλογο ερωτήσεων που θα πρέπει να απαντηθούν πριν ληφθούν κάποιες αποφάσεις πριν από τους επόμενους διαγωνισμούς προκηρύξεις και τα λοιπά προμηθειών. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν κάποιες απαντήσεις γιατί σαν παράδειγμα επιλέγεται στη μία περίπτωση η τάδε διαδικασία, γιατί εφαρμόζεται η διαδικασία αυτή με συγκεκριμένο τρόπο κτλ. Θα υπάρξει ένας κατάλογος με τα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί στο Κοινοβούλιο όπως το θέμα της ιδιοκτησίας, των οικοπαίδων επί των οποίων οικοδομούνται τα κτίρια, η ιδιοκτησία, η ενοικίαση των κτίριων, μακροπρόθεσμες ή βραχυπρόθεσμες μισθώσεις κτλ. 150 ερωτήσεις περίπου θα πρέπει να τύχουν απάντησης στην αρχή και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και όχι μόνο δύο εβδομάδες πριν πάρει τις αποφάσεις του το Κοινοβούλιο. Με τέτοιο τρόπο θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση, να αυξήσουμε τη διαφάνεια στην κτηριακή πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είμαι λοιπόν υπέρ του να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό επιτέλους και όπως σας είπα προσποθώ σε συνεργασία με άλλα μέλη της, της Επιτροπής μας θα καταλήξουμε σε μια διαδικασία ελπίζω ενδιαφέρουσα για όλους. Καλώς περνάμε στο επόμενο σημείο απαλλαγή 2008, άλλα όργανα, Συμβούλιο, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή, Περιφερειακή Επιτροπή, Επιτροπή Περιφερειών μάλλον κτλ. Κύριος Σαρνέσκι έχει το λόγο. Γεια σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Είναι τιμή μου που μπορώ να παρουσιάσω τις απόψεις μου σχετικά με την απαλλαγή για τα όργανα αυτά. Θα προσπαθήσω να συγκεντρώσω την προσοχή μου στα βασικά σημεία και να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Θα ξεκινήσω με μια γενικής φύσης παρατήρηση. Αν έθετε κάποιος το εξής ερώτημα, πώς μπορεί να αξιολογήσει κανείς με μία μόνο φράση την πολιτική, την δημοσιονομική των ευρωπαϊκών οργάνων. Ποια θα ήταν η απάντηση. Η απάντηση θα ήταν ότι πράγματι ε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ε, το τι έχει κάνει και η Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών και ε, ο Διαμεσολαβητής και όλα τα λεγόμενα ε, μικρότερα όργανα ή άλλα καλύτερα όργανα. Υπήρχαν στο παρελθόν αρκετά προβλήματα σαν παράδειγμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Παίρνω ένα παράδειγμα με, την, με τον εσικό, εσωτερικό έλεγχο για τις ε, διαδικασίες προμηθειών. Παρ' όλα αυτά έχουν υπάρξει βελτιώσεις, ε, έχουν υπάρξει κάποιες κινήσεις τις οποίες θα χαρακτήριζα ε, θα έλεγα ενθαρρυντικές. Θα πρέπει ίσως να κάνουμε όμως κάποιες διακρίσεις όταν μιλάμε για τα θέματα αυτά. Η δική μου ευθύνη, η δική μου αποστολή δεν είναι να προκαλέσω μια διοργανική κρίση σε καμία περίπτωση ή να θέσω σε αντιπαράθεση ε, τα ε, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί βασικό χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι η ενότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη αντίδραση για τα προβλήματα από πλευράς του Συμβουλίου. Θέλουμε να υπάρχει μια ξεκάθαρη ε, αντίδραση από πλευράς του Συμβουλίου όπως ακριβώς συμβαίνει και με τα υπόλοιπα όργανα. Το Συμβούλιο δεν έχει παρουσιάσει μια ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων όπως το έκαναν τα υπόλοιπα ε, θεσμικά όργανα. Το Συμβούλιο θα έλεγα κρύβεται πίσω από αυτό που έχουμε ονομάσει Συμφωνία Κυρίων. Αυτή η συμφωνία κυρίων βέβαια, αυτό το Gentleman's Agreement, αυτό το Gentleman's Agreement, ξέρετε ότι έχει συμφωνηθεί εδώ και μία τεσσαρακονταετία. Ήδη δηλαδή είναι ενισχύ από την δεκαετία του 70 κάτω από συνθήκες οι οποίες ήταν εντελώς διαφορετικές. Είναι ένα ενσταντανέ αν θέλετε αυτή η συμφωνία της κατάστασης που σοβούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε κοινή αγορά, δηλαδή το τι συνέβαινε το 1970. Γιορτάζουμε τα 40 χρόνια ε, αυτής της συμφωνίας κυρίων και περιμένουμε επιτέλους από πλευράς του Συμβουλίου κάτι το διαφορετικό. δεν σέβεται κάποιους κανόνες ε, το Συμβούλιο, ε, δεν ε, είναι υπόλογο θα έπρεπε να είναι σε σχέση με τα δημοσιονομικά και νομίζω ότι αυτή η συμφωνία κυρίων είναι θα έλεγα η αφορμή είναι ένα άλοθη ουσιαστικά. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται καλύτερα, είναι τέρος του Συμβουλίου ναι, το, το Κοινοβούλιο είναι εταίρος του Συμβουλίου, συνεργάζεται μαζί του, είναι αρμόδια επί του προϋπολογισμού αρχή, θέλει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στις σχέσεις ανάμεσα στα όργανα και στον τρόπο λειτουργίας των οργάνων αυτών. Νίχιλ Νόβιτσουψολ, Νομίζω ότι ε, δεν έχουμε λοιπόν ουδέν το, το κενόν υπό τον ήλιον, συνεπώς θα πρέπει το Συμβούλιο να αλλάξει άποψη. Δεν θα πρέπει σαν ένας μποξέρ που νιώθει αδυναμία να προσπαθεί συστηματικά αμυντικά να αποφεύγει τα χτυπήματα του αντιπάλου αλλά θα πρέπει να δώσει ε, απάντηση στο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι το minimum minimorum, είναι το ελάχιστον το οποίο θα πρέπει να κάνει σεβαστό το Συμβούλιο. Θα πρέπει να μας ενημερώσει για την πρόοδο που έχει επιτελέσει ή για την έλλειψη πρόοδου στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα πιστώσεων εκτός λογαριασμών σύμφωνα με τους προσανατολισμούς του εσωτερικού του ελεγκτή. Είναι σαφώς ότι θα πρέπει να επαληθεύονται σωστά οι αποδείξεις, τα τεκμήρια των δαπανών. Θα πρέπει επίσης να δημοσιεύονται όλες οι διοικητικές αποφάσεις και αυτό είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση γιατί οι αποφάσεις αυτές ε, χρησιμοποιούνται μερικές φορές σαν νομική βάση για θέσεις του προϋπολογισμού. Θα πρέπει επίσης να δίδονται στο Κοινοβούλιο και στην αρμόδια επιτροπή του οι ετήσιε ή η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 7 του δημοσιονομικού κανονισμού στον οποίο ε, αναφέρθηκα από πριν. Όπως ακριβώς δηλαδή κάνουν όλα τα υπόλοιπα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει από πλευράς του Συμβουλίου μία εξαντλητική ε, παρουσίαση των τεκμηρίων που απαιτούνται κάθε φορά όταν υπάρχουν μεταφορές ανάμεσα σε θέσεις του προϋπολογισμού. Και θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία τίθενται από τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι το οποίο μέχρι τώρα δυστυχώς δεν γίνεται και περιμένουμε εν πάση περιπτώσει από το Συμβούλιο ε, και τις προφορικές έστω εξηγήσεις στα ερωτηματικά του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Απαιτούνται σε πάρα πολλούς τομείς περαιτέρω θα έλεγα εξηγήσεις. Έχω εμείνει όπως βλέπετε στο Συμβούλιο γιατί έχουμε να κάνουμε με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία χρονίζουν σχετικά με το Συμβούλιο. Παρουσιάζει δηλαδή κάποια ιδιόρυθμα χαρακτηριστικά. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη κοινοβουλευτική πείρα και ίσως θα μπορούσαν να αναφερθούν και στο τι ακριβώς είχε συμβεί στο παρελθόν γύρω από την υπόθεση αυτή συμπληρώνοντας έτσι ε, την δική μου παρουσίαση. Τώρα να αναφερθώ πολύ συνοπτικά θα μου επιτρέψετε και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα με τα οποία ασχολήθηκα. Σχετικά με το ε, δικαστήριο, εδώ υποστηρίζω την άποψη του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με το δικαστήριο, την απαλλαγή. Κάνει ορισμένες συστάσεις στο ελεγκτικό συνέδριο προς το δικαστήριο σχετικά με τις ε, προμήθειες ε, κτλ. Έχεις. Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε την δημιουργία εσωτερικού ελέγχου στο δικαστήριο, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα θετικό και συγχαίρουμε το δικαστήριο. Για το ελεγκτικό συνέδριο δεν υπάρχουν προβλήματα και εδώ υπάρχει μια σύσταση θα έλεγα. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας ε, των δραστηριοτήτων του συνεδρίου θα πρέπει να υπάρχει μια πιο ε, ορθολογική δομή, διάρθρωση και καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ελεγκτικού συνεδρίου. Ένα τμήμα των θέσεων που υπάρχουν στο οργανόγραμμα ε, του ε, συνεδρίου πρέπει να γίνουν αντικείμενο διαχείρισης με πιο αποτελεσματικό τρόπο πέραν τούτου ουδέν για το ελεγκτικό συνέδριο για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή δεν έχουμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι σημαντικό να θυμίσουμε όμως την μεγάλη σημασία, το τεράστιο βάρος που έχει η συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή Περιφερειών και την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Αυτή η μορφή θεσμικής συνεργασίας και διοικητικής κυρίως συνεργασίας είναι σαφέστατα καλοδεχούμενοι. Τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειών θα πρέπει επίσης να καταθέτουν δηλώσεις ε, σχετικά με τα ίδια οικονομικά συμφέροντα έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαφάνεια την οποία όλοι επιδιώκουμε. Αλλά δεν υπάρχει κάποια περαιτέρω παρατήρηση. Πάντως πρέπει να γίνονται οι δηλώσεις αυτές όπως αυτή την οποία παρουσιάζουν οι ευρωβουλευτές εφόσον τις παρουσιάζουν οι ευρωβουλευτές, γιατί να μην είναι υποχρεωμένοι και τα μέλη της Επιτροπής των Περιφερειών να καταθέτουν ε, ε, αντίστοιχες δηλώσεις. Όλα αυτά θα έλεγα είναι επίπεδα διαφάνειας και ασφαλείας τα οποία ζητούνται, γίνονται αντικείμενο απέτησης από τον Ευρωπαίο πολίτη. Για τον διαμεσολαβητή δεν έχουμε επιφυλάξεις ε, σχετικά με την πρόταση που γίνεται. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μία τάση βέβαια στην αύξηση αν θέλετε του μεγέθους της υπηρεσίας, στην αύξηση της γραφειοκρατίας. Περάσαμε από 31 θέσεις στο οργανόγραμμα σε 57 αν δεν κάνω λάθος έχει ουσιαστικά υπάρξει ένας διπλασιασμός των θέσεων του οργάνου αυτού. Βέβαια εν μέρη υπάρχει και η τεκμηρίωση της αύξησης αυτής μέσω της αύξησης των αναφορών που κατατίθενται στον διαμεσολαβητή. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν έχουμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις θα πρέπει απλά να υπογραμμίσω μια σημαντική βελτίωση, θα έλεγα, στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αυτής της εξωτερικής υπηρεσίας. Υπάρχει μια σαφέστατη βελτίωση της λειτουργικότητας και του εσωτερικού συστήματος ελέγχου του συγκεκριμένου ε, οργάνου, υπηρεσίας καλύτερα αν θέλετε. Κλείνω, λέει ο κύριος Τσαρνέσκι, κύριε Πρόεδρε λέγοντας ότι υπάρχουν βελτιώσεις σε πολλούς τομείς. Υπάρχει όμως ένα σοβαρό πρόβλημα, υπάρχει ένα χένον πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που δεν θα μας οδηγήσει βέβαια σε μια βαθιά κρίση, αλλά υπάρχει ένα θέμα ανάμεσα στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Στην ουσία βιώνουμε εκ νέου καταστάσεις τις οποίες είχαμε συναντήσει και στο παρελθόν πριν 2-3 χρόνια. Εμείς ευχόμεθα να υπάρξει από πλευράς του Συμβουλίου μια μεγαλύτερη διάθεση συνεργασίας. Εμείς θέλουμε να υπάρχει εταιρική σχέση με το Συμβούλιο. Δεν είμαι θα αντίπαλοι του Συμβουλίου, είμαι θα εταίροι που σύμφωνα με τις αρμοδιότητές μας ελέγχουμε μέρος των δραστηριοτήτων του. Σήμερα το πρωί απεστάλησαν οι επιστολές προς την Προεδρία του Συμβουλίου. Περιμένουμε την απάντηση στις επιστολές αυτές. Και επαναλαμβάνω, εμείς δεν θέλουμε να υπάρξει μια θεσμική επανάσταση, θέλουμε απλά την βελτίωση του πραγματικού ελέγχου, αυτό αναμένει άλλωστε από εμά οι εκλογές μας. Σόντεμπεργκ. Tak formand. jeg deler generelt øh, øh de holdninger, som, øh, som øh, ligger Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις λεπτομέρειες τις οποίες μας έδωσε. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω κάποια μικρά σχόλια. Το πρώτο αφορά αν θέλετε το τυπικό του πράγματος. Έχει σημασία στην αρχή ενός τέτοιου ψηφίσματος να γίνεται αναφορά στα έγγραφα που υιοθετήσαμε τον Νοέμβριο ε, στις 23 Νοεμβρίου του 2009 με πολύ μεγάλη πλειοψηφία γιατί αυτή είναι η βάση θα έλεγα που μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα. Δεύτερον, αναφέρθηκε ο εισηγητής στη Συμφωνία Κυρίων στα σημεία 4, 5 και 8. Κατανοώ ότι πέρυσι στα πλαίσια της συζήτησης είχαμε πει ότι δεν θα θίξουμε το θέμα της συμφωνίας κυρίων. Γιατί αναρωτιόμασταν τι είδου συμφωνία είναι αυτή, δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι. Θα ζητήσαμε ένα έγγραφο το οποίο να αναφέρεται στη συμφωνία αυτή, επίσημο, δεν πήραμε τίποτα. Και γι' αυτό παρακαλώ να επανέλθουμε σε αυτό που είχαμε αποφασίσει πέρυσι αν υπάρχουν βέβαια οι οποίοι θέλουν, αυτοί που θέλουν να, συμπεριλάβουμε τη συμφωνία των κυρίων αυτοί, τότε να παρουσιαστεί, να κατατεθεί στα έγγραφα έτσι ώστε να ξέρουμε ακριβώς με τι έχουμε να κάνουμε. Μιας και όμως αναφερόμαστε συνεχώς σε κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, τότε χάνουμε το χρόνο μας. Και νομίζω ότι η περσινή μας απόφαση ήταν και παραμένει σωστή. Και θα ήθελα το ίδιο ακριβώς να κάνουμε και φέτος. Το τρίτο σημείο στο οποίο θα σταθώ αφορά το σημείο 11. Ίσως εδώ να υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα μεταφραστικό περισσότερο. Νομίζω όμως ότι η διατύπωση ως έχει δεν είναι πάρα πολύ ε, θα έλεγα ικανοποιητική, τουλάχιστον στην γλώσσα στην, ε, στα Δανέζικα. Εμείς, εμείς θέλουμε το Συμβούλιο όχι να λάβει υπόψη τις ερωτήσεις μας, όχι να υπενθυμίσουμε στο Συμβούλιο τις ερωτήσεις που έχουμε επανειλημμένα θέσει στη διάρκεια του χρόνου, αλλά να δώσει απαντήσεις στο Συμβούλιο ή έστω να προσπαθήσει να απαντήσει το Συμβούλιο στις ερωτήσεις αυτές. Σαν παράδειγμα, οι υπηρεσίες οι εκτός προϋπολογισμού αναβαπτίστησαν από ό,τι βλέπω. Άλλαξε εντελώς η ονοματολογία. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι αυτό συνιστά απάντηση στις ερωτήσεις τις οποίες θέσαμε για τις υπηρεσίες αυτές εκτός προϋπολογισμού. Τέταρτο, Έχω την αίσθηση ότι όταν δει κανείς το τι συνέβη πέρυσι και όταν απλά θέλει κάποιος να ενημερώσει λίγο την κατάσταση, να δει τι συνέχεια υπάρχει, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν αυτά παραδείγματα στον τρέχοντα προϋπολογισμό που να περιγράφουν την κατάσταση πάρα πολύ καλά. Θυμίζω ότι στους λογαριασμούς του 2009 υπήρχαν τεράστια ποσά, εκατομμύρια ε, ευρώ που πήραν ας πούμε ε, και πήγαν από το κεφάλαιο της Γερμηνίας στο κεφάλαιο των διοικητικών δαπανών γενικότερα και μετετράπηκε η φύση των δαπανών αυτών, των πιστώσεων αυτών. Αναρωτιέμαι τι συνέβη το 2008. Η πρακτική αυτή η οποία μας προκάλεσε το 2007 συνεχίστηκε Μας ζήτησε, προσπάθησε το Συμβούλιο να ακούσει τις προσπάθειες, τις προσπάθειές μας, ε, τις συστάσεις μας ή μήπως μας αγνόησε όπως διαπιστώσαμε ότι μας είχε αγνοήσει και πέρυσι. Το Συμβούλιο είναι παρόν εδώ σήμερα, ε, μπορεί ίσως να δώσει κάποιες απαντήσεις. Επαναλαμβάνω, συστηματικά επιθυμία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα στενότερος διάλογος με το Συμβούλιο. Ο διάλογος αυτός θα φέρει στην επικαιρότητα τις βελτιώσεις όποιες και αν είναι αυτές εφόσον έχουν συμβεί. Τέλος, αυτό που θα ήθελα να μάθω πριν από την επόμενη συνάντηση από τον εισηγητή και τον πρόεδρο να προσκαλέσουν το Συμβούλιο σε μία επίσημη αντιπαράθεση, επίσημη συζήτηση έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτηματικά που θέτουμε. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι την προσπάθεια αυτή την έχουμε ήδη κάνει. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση και είναι σαφές ότι σύντομα θα πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση με το Συμβούλιο. Ο κύριος Ριβελίνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί και με αποφασιστικό τρόπο και χρησιμοποιώντας θα έλεγα μια συμπαθητική αλλά αποφασιστική γλώσσα έφερε στην επικαιρότητα μια σειρά προβλημάτων σοβαρών. Τα προβλήματα αυτά έχει φτάσει η ώρα να επιληθούν. Εάν δεν το κάνουμε αυτό σήμερα και απλά δώσουμε για μια ακόμη φορά την σύμφωνη γνώμη μας, πότε θα το κάνουμε. Έχουμε την δυνατότητα να επηρεάσουμε κάποια προβλήματα έτσι ώστε να επιληθούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από το 1970 έχει αλλάξει. Δεν έχει καμία σχέση η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το οποίο προϋπήρχε στη δεκαετία του 70. Ο κόσμος έχει αλλάξει εντελώς. Κάποιες συμφωνίες κυρίων που ήταν καλές για το 1970, ε, οι συμφωνίες αυτές είναι άχρηστες, εντελώς περιτές σήμερα. Συνεπάς, συνεπώς, ή, ε, σχετικά με το Συμβούλιο, δεν θα πρέπει να δώσουμε την απαλλαγή πλέον. Θα πρέπει να αρνηθούμε την απαλλαγή προς το Συμβούλιο. Θα πρέπει να επανεξετάσουμε αυτές τις περίφημες συμφωνίες του 1970 και υπάρχει πλέον η δυνατότητα για την πλήρη αναθεώρηση της σχέσης μας με το Συμβούλιο. Ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου πλέον συνάδελφοι θα διαχειρίζεται πιστώσεις πολύ ψηλότερες από ό,τι στο παρελθόν. Συνεπώς έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή την ευκαιρία να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με το πρόβλημα. Για το δικαστήριο. Ο εισηγητής ε, μας ε, σημειώνει μία σειρά από αδυναμίες. Ε, καταρχάς η μονογλωσία σε ορισμένες δραστηριότητες του δικαστηρίου, όπως επίσης και οι προκηρύξεις για προμήθειες κτλ. Ε, νομίζω ότι οι παρατηρήσεις τις οποίες κάνει ο εισηγητής δείχνουν ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται από το δικαστήριο είναι πολύ ατελείς. Θα πρέπει λοιπόν να φανούμε προσεκτικοί αλλά παρόλα αυτά να χορηγήσουμε την απαλλαγή. Δεν λέω ότι δεν θα ήταν σωστό το να μην χορηγήσουμε την απαλλαγή αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι καλό θα είναι η Επιτροπή μας να την χορηγήσει. Για το ελεγκτικό συνέδριο υπάρχει ένα θέμα. Για μένα υπάρχει ένα θέμα το οποίο κρίνω πάρα πολύ καθοριστικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει μια έλλειψη θα έλεγα καλή συμπεριφοράς απέναντί μας όταν ανακοινώνει, παρουσιάζει το συνέδριο τις εκθέσεις του, τις ειδικέ εκθέσεις πρώτα στον τύπο και μετά σε μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνω απαράδεκτο. Είναι αδικαιολόγητο και θα πρέπει να αναθεωρηθούν θέματα τα οποία είναι μεν σε ένα πρώτο επίπεδο, τυπικά θέματα αλλά ε, μετατρέπονται σε θέματα ουσίας εκ των υστέρων. Θα πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε ότι εδώ είμαστε ε, εκπρόσωποι των λαών της Ευρώπης και δεν πρέπει να μας αγνοούν. Είναι σαφές ότι αυτό το θέμα το συνέδριο θα πρέπει να το ελέγξει πολύ καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Έχει δίκιο η συγκητής όταν ζητά επίσης και την κατάθεση των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του ε, συνεδρίου όπως επίσης και του δικαστηρίου. Σύμφωνο επίσης και με την στρατηγική ε, του ελεγκτικού συνεδρίου σε επίπεδο διαχείρισης ε, του ανθρώπινου δυναμικού. Τώρα για τον προϋπολογισμό της Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Νομίζω ότι μιλάμε για εκλεγόμενα μέλη. Συνεπώς οι καταθέσεις δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων της, ε, των μελών της ΕΚΟΣΟΚ, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής είναι απαραίτητη. Για τα θέματα ε, του διαμεσολαβητή υπάρχουν κάποιες απορίες τις οποίες διευκρινίζει πολύ ο κύριος Τσαρνέσκι δεν υπάρχει θέμα να μην χορηγήσουμε την απαλλαγή. Το ίδιο ισχύει επίσης και για την υπηρεσία δεδομένων, προσωπικών δεδομένων. Τελειώνω. Επαναλαμβάνοντας, υπενθυμίζοντας αυτά τα οποία σας είπα στην αρχή, έχει φτάσει η στιγμή έτσι ώστε να διευκρινιστούν ορισμένες καταστάσεις. Αν δεν διευκρινιστούν τώρα δεν θα έχουμε καταλληλότερη στιγμή. Πρέπει να το κάνουμε τώρα γιατί είναι καθήκον μας να διαλυθούν προβλήματα τα οποία χρονίζουν. Ευχαριστώ τον Σαργέσκη για την προσπάθεια την οποία έκανε και για τη γλώσσα την οποία χρησιμοποίησε αποτελεσματική, σκληρή σε εισαγωγικά, αλλά κυρίως επαναλαμβάνω αποτελεσματική. Βέλεα. Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Συμφωνώ επίσης με όσα είπε και με τα όσα σχολίασαν οι προηγούμενοι δύο α, συνάδελφοι που νομίζω ότι ήταν αυστηροί αλλά προσεκτικοί στις διατυπώσεις τους. Πάντως όλα αυτά είναι γνωστά ακόμα και όσον αφορά τις επικρίσεις προς το Συμβούλιο γιατί τα ίδια λέμε κάθε χρόνο. Μερικά λάθη είναι ασυγχώρητα. Ε, του λένε παράδειγμα προς μίμηση για τα άλλα θεσμικά όργανα. Επίσης, φυσικά και είναι υψηλό το ποσοστό λαθών και από εθνικές ε, αρχές για άλλη μια φορά. Το Συμβούλιο βέβαια δεν ήρθε στην ε, συνάντηση. Ενώ το Συμβούλιο θα έπρεπε να είναι φίλος συνεργάτης, θα έπρεπε ε, να υπάρχει επικοδημητικό πνεύμα στις σχέσεις μας. Και οπότε την ώρα που κρίνεται η απαλλαγή και έγκριση του προπολογισμού, τότε, τότε, τότε δείχνει πνεύμα συνεργασία. Όμως δεν καταλαβαίνω γιατί τώρα εν προκειμένου ε, δεν, δεν, δεν, δεν ε, έρχεται στην παρούσα συζήτηση. Τι γίνεται ε, όταν ε, κάτι έχει να κάνει με την τσέπη μας τότε ζοριζόμαστε. Έχουμε το θέμα της Λισαβόνας, διότι τώρα θα γίνει με ισχύουσα τη συνθήκη η έγκριση της οικονομικής διαχείρισης. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς το Συμβούλιο θα τοποθετηθεί, πώς θα απαντήσει σε όλα αυτά τα οποία ανακύπτουν. Όλα αυτά τα οποία έχει θέσει εύστοχο ο κ. Τσαρνέτσκι που μας είπε ότι η στάση του Συμβουλίου μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ ε, χαλαρή. Προσοχή όμως γιατί τώρα έχει αρχίσει μια καινούργια διαδρομή, μια καινούργια εποχή. Άρχισε να ισχύει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα πρέπει ομένω το Συμβούλιο να δείξει μεγαλύτερη πρωτοβουλία. Θα πρέπει να μα πει τι πρεσβεύει. Έχω μια ερώτηση για τον ε, εισηγητή. Τι, τι, τι γίνεται, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σχέση μας με το Συμβουλίο. Πού είναι οι απαντήσεις του Συμβουλίου, δεν υπάρχουν πουθενά. Τι διαδικασίες ισχύζουν. Εγώ θεώρησα ότι έχει γίνει βήμα πρόοδο την τελευταία ώρα που τα είπαμε. Άρα, εάν δεν είσαι κάτι να ξέρουμε τι γίνεται. Θα πρέπει και η Προεδρία να εμπλακεί στη διαδικασία της απαλλαγής. Μα τι γίνεται εδώ, αγνοείται η νομιμότητα από πλευράς του Συμβουλίο. Για να το κοιτάξουν αυτό παρακαλώ οι συγγητές μας. Κάτι άλλο τώρα όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Η πρικοδότηση αλλά και το προσωπικό έχει αυξηθεί να κάνουμε όμως και να εξετάσουμε τι γίνεται, πώς η συγκυρία δικαιολογεί μια τέτοια αύξηση δαπανών σε αυτή την ε, υπηρεσία. Τώρα στον αυτό συνέδριο θα πρέπει να προσέξουμε κάτι το οποίο το ξεχνάμε καμιά φορά που είναι ε, η δημοσίευση των ε, οικονομικών συμφερόντων. Θα πρέπει και αυτό ε, στο βωμό της ε, διαφάνειας να ανέβει στο ίντερνετ. Και για την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επίσης να δούμε κατά πόσον μπορούμε να υπολογίσουμε τα αποτελέσματα ε, της συνεργασίας με αυτό το θεσμικό όργανο με τρόπο συγκεκριμένο. Αντρέασεν. Η έκθεση του κ με ανησυχεί. Σα επισήρω Σας την προσοχή. Προσοχή, προσοχή όσον αφορά την απαλλαγή. Εγώ έλεγα όχι, τελικά δόθηκε το πράσινο φως στο Συμβούλιο τον Νοέμβριο. Very grateful for this report from Mr. Czarnesky. I find it Τελικά μετά από όλα αυτά όμω, νομίζω ότι παρά είναι ε, ποιητή ο κύριο ε, Τσανεσκινά στο, στο, στο 11. Όχι, πέρασε η εποχή των ερωτήσεων. Τώρα ήρθε η ώρα τη διαπίστωση του αν όσα είπαμε σαν προπόθεση απαλλαγή, αν ισχύουν. Για παράδειγμα, τι έγινε με, με, με, με τα ε, κονδύλια του προπολογισμού τα, τα έκτακτα. Αυτά δηλαδή που ζητήσαμε πέρσι γίνανε. Αλλιώς δεν δίνουμε την απαλλαγή. Τη δώσαμε τον Νοέμβριο επί τη βάση του ότι θα συμμορφωθούν με τα όσα ζητήσαμε. Άρα δεν είναι η ώρα των συναντήσεων και των ερωτήσεων. Είναι η ώρα της διαπίστωσης αν κάνανε αυτά που έπρεπε. Βασικά συμφωνώ από με τον κύριο Ριβελίνη. Να αναλάβουμε δράση. Τέρμα η αναμονία. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στον συνάδελφο για το Συμβούλιο και πέρσι αρμόδιος ήταν ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος θα πρέπει να έρθει. Ή τέλο πάντων όποιο είναι είτε στον ειναι η προεδρια κάποιος να έρθει. Να ξεκαθαριστεί το εάν τα λέμε σωστά. για τους αποδέκτες. Γιατί πέρσι ήταν σαφές ότι ο συνομιλητής μας ήταν ο Γενικός Γραμματέας. Τι έγινε από πλευράς Προεδρίας. Έχει λάβει τη λίστα των ερωτημάτων μας. Ή όχι η Προεδρία. Να μας πει ο εισηγητής. Να μας δώσει και ένα αντίγραφο των όσων απίθυνε στην Προεδρία. Ποιο είναι ο συνομιλητής μα, Ποιο είναι ο υπεύθυνο για αυτά που ζητήσαμε να κάνει το Συμβούλιο. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή, ο κύριος Σαρμάς από πλευράς ε, του ελεγκτικού συνεδρίου έχει το λόγο. Δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, λέει εκπρόσωπο του συνεδρίου. Ο εισηγητής κ. Τσανέσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, τους εκλεκτούς συναδέλφους για τις παρατηρήσεις τις οποίες έκαναν. Τις βρήκα όλες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και τον προκάτοχό μου για την έκθεση που είχε κάνει και την οποία εν πολλής χρησιμοποίησα. Εγώ φυσικά αντιτίθεμαι πλήρως σε σχέση με αυτή τη συμφωνία κυρίων. Νομίζω για τον κύριο Σέντεργαρντ, όπως και η κυρία να αναγνωρίζουν ότι είναι σοβαρό το θέμα. Ίσως η διατύπωσή μου να ήταν ιδιαίτερος soft και διπλωματική στο σημείο 11. Αλλά είναι αλήθεια ότι προσπάθησα να είμαι απλά πολύ ευγενής, τίποτα περισσότερο. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ βρισκόμαστε να καταθέτουμε για μια ακόμη φορά, για δεύτερη, τρίτη φορά, τις ίδιες ερωτήσεις. Αυτό αποδεικνύει ότι το Συμβούλιο στον ενδιάμεσο χρόνο δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Οι παρατηρήσεις τις οποίες έκανε επίσης ο κύριος Ριβελίνη είναι πολύ σωστές. Είναι σαφές ότι η δεκαετία του 70 είναι πάρα πολύ μακριά και πίσω μας. Σχετικά με το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει υπάρξει πρόοδος. Παραδεχόμαστε την πρόοδο αυτή και χορηγούμε την απαλλαγή για το ελεγκτικό συνέδριο. Έχει τεθεί ένα σοβαρό πρόβλημα βέβαια Νομίζω ότι αυτό δείχνει την ποιότητα της συζήτηση που είχαμε στις αρχές του φθινοπόρου στην Επιτροπή μας. Πράγματι τότε είχε ενημερωθεί πρώτα ο τύπος από το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι θέμα, αν θέλετε, ύφους, είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Στα πολωνικά τι λέμε. Λέμε ότι δύο πράγματα έχει κανείς να περηφανεύεται για την παιδική του ηλικία και για το σπίτι του. Τα ωραία του έπιπλα ή τον σωστό τρόπο με τον οποίο έχει ανατραφεί. Νομίζω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το ελεγκτικό συνέδριο επέλεξε τα έπιπλα. Λοιπόν, ο κύριος Ριβελίνη έχει δίκιο που έθεσε λοιπόν για μια ακόμη φορά το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ επίσης και την Βάιλα. Είπε πάρα πολύ σωστά ότι το Συμβούλιο θεωρητικά θα πρέπει να λειτουργεί σαν υπόδειγμα για τα υπόλοιπα όργανα και για τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βάιλερ, έχετε απόλυτο δίκιο και θα το χρησιμοποιώ αυτό πολύ στο μέλλον. Τώρα η πρόταση ε, για μια επίσημη, ανεπίσημη, διμερή συνάντηση με το Συμβούλιο. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ. Σχετικά με την παρατήρηση της κυρίας Γκρέσλερ. Βρισκόμαστε σε μια στασιμότητα κυρία Γκρέσλε. Δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικές ποιοτικέ βελτιώσεις, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος σχετικά με το Συμβούλιο και τη στάση του. Ευχαριστώ την κυρία Γκρέσλα για τις προτάσεις της και για τις συστάσεις της έτσι ώστε να ελέγξουμε τις αυξήσεις ε, που έχουν απαιτηθεί και για τον ε, διαμεσολαβητή και για ε, την υπηρεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και σε ποιο βαθμό οι αυξήσεις αυτές του οργανογράμματος βελτιώνουν τη λειτουργία τους. Τώρα σχετικά με την δήλωση οικονομικών συμφερόντων και του ελεγκτικού συνεδρίου είναι μια ιστορία η οποία επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται συνεχώς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να υπενθυμίσουμε ακριβώς και στα πλαίσια της διαδικασίας για το διορισμό των νέων μελών του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ και την κυρία Άντρεασεν. Πράγματι ασκεί κριτική στις ρυθμίσεις τις οποίες εγώ απλά σχολίασα και εν πολλής συμπληρώνει αυτά τα οποία είπα εγώ και την ευχαριστώ γι' αυτό. Θυμίζω ότι το σημείο 11 πρέπει να είναι ίσως λίγο πιο σκληρό αν θέλετε, αλλά προσπαθώ να κρατήσω την ε, ψυχραιμία μου. Εγώ δεν χάνω την ψυχραιμία μου εύκολα. Ε, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να χάσω την ψυχραιμία αυτή. Για την κυρία Αγιάλα Σεντέρ νομίζω ένα πράγμα θα πρέπει να θυμίσω. Ήσασταν η πρώτη Ευρωβουλευτής, κυρία Αγιάλα Σεντέρ, που συνάντησα πριν πέντε χρόνια όταν μπήκα μέσα στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το θυμάμαι πάντα, η συνάντησή μας με έχει σημαδέψει κυρία Ιάλα Σεντέρ. Έχει υπάρξει λοιπόν πρόταση για συνάντηση με το Συμβούλιο και σας ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Σας ευχαριστώ και εγώ όλους για όλες τις διαδικασίες απαλλαγής. Η προθεσμία είναι η Παρασκευή 2 Μαρτίου. Περνάμε στο τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Απαλλαγή για το 7ο, 8ο και 9ο πρόγραμμα, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξη. Δίνω το λόγο στην κυρία Αγιάλα Σέντερ, η συγγήτρια. Sí, gracias. Perdone, voy a mirar dónde tengo los documentos, que no sé dónde los he perdido. En el, ah, sí, en el viaje. Ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε να βρω τα έγγραφά μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα θα ευχαριστήσω τις και τους συναδέλφους για την ενδιαφέρον που έριξαν για να συζητήσουμε. Ευχαριστώ και για τις τροπολογίες, ήδη από τώρα, τις οποίες θα καταθέσετε. Συναντήθηκα κατά επανάληψη με τον κύριο Κίβιτς, με τους εκπροσώπους της Κομισιόν. Όλα αυτά οδήγησαν σε ανταλλαγές απόψεων. Συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εξετάζουμε πού μπορεί κανείς να επιτύχει κάποιος πρόοδους και πού χρειάζεται να επιτύχουμε κάποιες βελτιώσεις. Ο κ. Ουκιέβιτς είπε ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν περιληφθεί εννοώ δηλαδή τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου, εδώ πρόκειται για τον μελλοντικό πολιετή δημοσιονομικό σχεδιασμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αναπτύξεως θα πρέπει να ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Ένωσης και να μην εξαρτάται από ειδικά από ειδικέ διατάξεις. Να μπει εκεί και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, γιατί όπως είναι τώρα οι ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα περίπλοκες. ο νέος πολιετής σχεδιασμός θα γίνει στη βάση της συνθήκης της Λισαβόνας, θα υπάρξει μια αναδιάρθρωση. Ορισμένες αμφιβολίες που έχουμε σχετικά με το μελλοντικό πολιετή σχεδιασμό υπάρχει και ένα μεγάλο ε, ένας μεγάλος άγνωστος που είναι η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία εκεί πρέπει να σκεφτούμε κάπως ποια θα είναι η μελλοντική διάρθρωση πρέπει να ρίξουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένους τομείς που θεωρήσαμε ότι είναι πλέον σημαντικοί και πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι μη κρατικές οργανώσεις να μην υποστούν αυτές δυσμενείς επιπτώσεις γιατί αυτές είναι που εργάζονται επί τόπου ίσως βέβαια υπάρχουν κάπως υπερβολικά πολλές μη κρατικές οργανώσεις αλλά αυτό δεν επιτρέπεται να, να καταλήξει στο να μην μπορούν οι σημαντικές ε, μη κρατικέ οργανώσεις να απευθύνονται σε εμά και να λαμβάνουν βοήθεια. Γιατί όπως είπα αυτές είναι οι οποίες ε, ε δραστηριοποιούνται επί τόπου όταν, όπου υπάρχει ανάγκη. Άλλα θέματα που έχω συζητήσει και με το ελεγκτικό συνέδριο και που μας ανησυχούν είναι το περιθώριο, ε, τα ποσοστά ασφάλματος μάλλον, σημειώθηκε μια σειρά σφαλμάτων στις πληρωμές που δεν είναι δυνατόν πάντοτε να ποσοτικοποιηθούν σε ό,τι αφορά τις διάφορες ε, βοήθειες. Ε, ως Επιτροπή ζητούμε από την Κομισιόν να μας προτείνει μηχανισμούς και συστήματα που θα καταστήσουν δυνατόν να αντιμετωπιστεί αυτός ο κατακαιρματισμός των διατάξεων ώστε να βελτιωθούν τα υφιστάμενα συστήματα. Η Κομισιόν ήδη από θα το πράξει αυτό, ώστε να μειωθεί το ποσοστό των σφαλμάτων. Δύο άλλα θέματα τώρα. Εξών το ένα έχει σχέση με τις δημοσιονομικές βοήθειες. Κυρίως άμεσες βοήθειες όταν σημειώνονται κρίσεις σε ορισμένες χώρες βλέπε Αγγόλα στο παρελθόν επίσης στην Αϊτή στον Νίγηρα ενδεχομένως άμεσες βοήθειες από τον προϋπολογισμό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Αναπτύξεως ή από άλλα ταμεία πρέπει να δούμε εκεί πώς θα λειτουργήσουν οι μηχανισμοί ελέγχου αν είναι δυνατόν να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ερωτήσεις αυτές, γιατί υπάρχει ήδη παρά την Κομισιόν ένα σύστημα χορήγησης άμεσης βοήθειας όταν ε, ε, συμβαίνει κάποια θεομηνία, όταν ε, σε κάποια χώρα αρχίζει ένας πόλεμος ή ένας εμφύλιος πόλεμος ή τέλο πάντων όταν υπάρχει μια εκτεκτή ανάγκη. Το όλο πλαίσιο γίνεται πιο περίπλοκο τώρα και δεν είναι και τόσο ε, διαφανές. Τα λέω αυτά στην έκθεσή μου. Μαζί με το ελεγκτικό Συνέδριο θα χρειαστεί να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να εγγυάται μια απλοποίηση και βελτίωση των ελέγχων σε, αυτούς, σε αυτές τις πληρωμές επίγοντος χαρακτήρα. Εδώ είναι σαφές ότι το ελεγκτικό συνέδριο δεν μπόρεσε να ελέγξει τις ε, ε, Συναλλαγέ αυτές, ότι δεν υπήρχαν σχετικά έγγραφα. Και με αυτά τα παραστατικά επομένως μπορέσε να γίνει η κρίση και άρα θα πρέπει και η Κομισιόν να κατεβάσει κάποιες προτάσεις. Ότι δηλαδή εάν για τις ε, τρέχουσες και κατεβίουσες συναλλαγές ισχύει ένα σύστημα, εάν είναι αρκετά αποτελεσματικό, κάτι το οποίο δεν συμβαδίζει με την κρίση του ελεγκτικού συνεδρίου. γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλες για, όλα τα, τα, θεσμικά όργανα και μίλαγα με τον κύριο Ντεχίχτ και λέγαμε για τον ΟΗΕ ότι εκεί δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα παραστατικά την, την ώρα που γινόταν ο οικονομικός έλεγχος και μου είπε ότι αντίθετα η Κομισιόν έχει τα αντίστοιχα έγγραφα αλλά δεν τα έχει δώσει στο συνέδριο. Για να μας πούν τι ισχύει. Οπότε... Για διάφορες υπηρεσίες, όπου την υπηρεσία συγκρότησης του κοσυφοπαίδιου κλπ. Θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται. Τι ισχύει, γιατί έχουμε τις εξωτερικές μας πολυμερείς σχέσεις που έχουν κάποιο παρελθόν. Συμφωνούμε σε πολιτικό επίπεδο. Θέλουμε αυτή την, την πολυμερή συνεργασία με ΟΗΕ και άλλους, αλλά, αλλά από πλευράς ε, οικονομικού ελέγχου ισχύουν άλλα. Πώς γίνεται ο έλεγχος. Ο καθένας έχει άλλο σύστημα ελέγχου. να υπάρχει διαφάνεια. Μπόρεσε το συνέδριο να κάτσει και να ζυγίσει και να μετρήσει το τι γίνεται κατά τις σχέσεις μας και συναλλαγές μας με αυτούς τους οργανισμούς. Τώρα, για τους ανθρώπινους πόρους. Είπα αυτή την ε, συγκυρία οπότε και διαμορφώνεται ένας νέος ρόλος στην διεθνή σκηνή για την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι βγήκαμε μπροστά πρωτοπόροι όπως και για την τραγωδία της ΑΕΤΗΣ η Ένωση μέσω της Κομισιόν και ο ΙΕ Οπότε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας για ασφάλεια, σταθερότητα και αποτελεσματική χρήση των ανθρωπίνων πόρων. Άρα και σε αυτό το επίπεδο να μας πει η Κομισιόν. Τι προτάσεις έχει. Τι μπορεί να κάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου για την καλύτερη αξιοποίηση των ανθρωπίνων πόρων. Να πιάνει τόπο το προσωπικό που διαθέτουμε. Γιατί να πρέπει να δούμε και τη γίνεται και σχετικά με τα αιτήματα που έχει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Περιμένουμε επομένω την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα τα ξαναπούμε πάντως, δεν θα κλείσει σήμερα το θέμα. Οπότε δύο του Πρόεδρου ελπίζω να διαφωτιστούμε στα πλαίσια αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πρώτα την ε, κυρία συνάδελφο, την κυρία Αγιάλα Σέντερ, για την θετική συνεργασία. Βεβαίως και η έκθεση μου φαίνεται διατυπωμένη με ακρίβεια και ότι αποδίδει τα σημαντικότερα θέματα. που μας απασχολούν σχετικά με την περιφερειακή, με την αναπτυξιακή βοήθεια μάλλον. Δυστυχώς και στο μέλλον φαίνεται η αναπτυξιακή βοήθεια να είναι κατακαιρματισμένη εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και στο μέλλον λοιπόν θα έχουμε ανάγκη να ζητούμε μια πολιτική με ιδιαίτερα στοχευμένη από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώ μέσα στην Κομισιόν δεν υπάρχουν οι αναλογούσες δομές ώστε να μπορέσει να κινηθεί η υπόθεση αυτή προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Δεύτερο, τονίζω ότι και όταν θα δημιουργηθεί η εξωτερική υπηρεσία πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς κατά πόσον η αναπτυξιακή βοήθεια θα διαλαμβάνεται μεταξύ των στόχων της υπηρεσίας αυτής και ούτω καθεξής, θα είναι ο ρόλος της ε, πολιτικής γειτονίας Δηλαδή, με ποιον τρόπο θα γίνει ένας πραγματικός αποτελεσματικός συντονισμός με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να μιλεί κανείς για μια στοχευμένη πολιτική. Εν προκειμένου τονίσω ότι διεξάγουμε και πολλές συζητήσεις περί προσφύγων, περί πολιτικής ασύλου που έχουν άμεση σχέση με το συζητούμενο θέμα. Διότι η αποτελεσματικότητα των αναπτυξιακών βοηθειών μπορούν να συμβά, μπορεί να συμβάλλει ώστε οι ε, άνθρωποι να δουν ότι έχουν κάποια πιθανότητα να ε, δράσουν οικονομικά στην πατρίδα τους και να μην χρειάζεται να την εγκαταλείψουν. Θα θίξω ιδίω δύο θέματα. Πρώτα τις δημοσιονομικές βοήθειες λέγοντας αυτό που είπε η Αγιά Σέντερ ότι δεν είναι ικανοποιητικό ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζονται. Ούτε το ελεγκτικό συνέδριο δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα για να αξιολογήσει τις πληρωμές αυτές. Και εκτός αυτού που περιέχονται και λάθη που δεν ήταν δυνατόν να ποσοτικοποιηθούν, πρόφανως και οι στόχοι που συνδέονταν με τις δημοσιονομικές αυτές βοήθειες δεν είχαν δεν μπόρεσαν να ελεγχθούν δεν υπήρχαν ούτε καν προϋποθέσεις δεν υπάρχει δηλαδή ένας συγκεκριμένο κατάλογος που να λέει με ποιον τρόπο και για ποιο λόγο δίνεται δημοσιονομική βοήθεια και τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνονται με ένα τέτοιο τρόπο που να βλέπει και ο Ευρωπαίος πολίτης ότι έχουν κάποιο νόημα. Όσο όλοι γνωρίζουμε, δυστυχώς σε ορισμένες από τις χώρες αποδέκτριες οι κυβερνητικές δομές είναι τόσο διεφθαρμένες όπου πραγματικά πρέπει κανείς να σκεφτεί εάν όντω οι δημοσιονομικές βοήθειες και η αύξησή τους είναι πραγματικά τόσο απαραίτητες και εύκολες όπως φαίνεται να προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θεωρώ ότι όχι. Τώρα, παράγραφος 35. Το investment facility. Συμφωνώ με την άποψη ότι εδώ στο Ευρωκοινοβουλίο πρέπει να ελέγξουμε με βοήθεια και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα προγράμματα πιστώσεων. Δηλαδή πραγματικά αποδίδουν στην επίτευξη των στόχων τους υπάρχει και μια ασάφεια. Λέμε ότι θέλουμε να βάλουμε το investment facility στην απαλλαγή. Δεν είναι όμως δικό μας καθήκον να ελέγξουμε εάν η συγκεκριμένη πίστοση δαπανήθηκε με το σωστό τρόπο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το πράξει η τραπεζική εποπτεία. δεν μπορεί να είναι καθήκον των κοινοβουλευτικών να διεξάγουν τραπεζική εποπτεία. Το ζήτημα που ενδιαφέρει είναι εάν οι πολιτικοί ουσιώδεις στόχοι έχουν επιτευθεί. Αυτά θα ήθελα να τα διαχωρίσω, διότι δεν έχουμε την εποπτεία των τραπεζών εμείς ως κοινοβουλευτικοί. Ευχαριστώ εν τέλει και το ελεγκτικό συνέδριο για την εξαιρετική συνεργασία. Παραλίγο λίγο να το λησμονήσω, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου, ο κ. Σούρτσνιεβίτς, εφόσον θέλει, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε το λόγο. Η πιο σημαντική ερώτηση την οποία έθεσε η κυρία Σέντερ είναι η εξής. Ζητά να υπάρξουν κάποιες προτάσεις οι οποίες να γίνουν σεβαστές. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι οι προτάσεις αυτές και το λέω με θετικό πνεύμα, υποστηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα όποια προβλήματα το ελεγκτικό συνέδριο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος εδώ. Θα πω ότι οι συστάσεις του Κοινοβουλίου είναι πλήρεις, ασχολούνται με τα σημαντικά προβλήματα, σχετικά με τα στοιχεία τα οποία ενημερώνεται το ελεγκτικό συνέδριο. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε βέβαια αν το ελεγκτικό συνέδριο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία μιας ομάδας διοργανικής εργασίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών των διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών ελέγχου, ελεγκτικών δηλαδή συστημάτων στο εσωτερικό ε, των μεγάλων οργάνων. Αυτό είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει πάρα πολλές δυσκολίες σε περιπτώσεις ε, επιδοτήσεων, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξει συνεργασία με όλα τα ελεγκτικά όργανα έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματικός τρόπος με τον οποίο ε, θα συνεχιστεί η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τις δωρήτριες χώρες. Ελπίζω ότι η κατάληξη των εργασιών αυτής της ομάδας θα μας οδηγήσει σε μια ουσιαστική απλούστευση. Ο εξωτερικός ε, θα έλεγα ελεγκτής θα έχει αποτύχει εφόσον δεν έχει θέση στη διάθεση των ενδιαφερομένων όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση. δεν είχαμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε ε, περισσότερο από ένα μικρό τμήμα του προϋπολογισμού γιατί δεν είχαμε τα απαραίτητα τεκμήρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω γενικότερα πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας έχει υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις δραστηριότητες τις οποίες έχουμε κάνει και οι οποίες έχουν σαν στόχο μια μεγαλύτερη διαφάνεια για αυτήν τη νέα μέθοδο βοήθειας η οποία προσφέρεται προς τρίτες χώρες. Ε, φυσικά και το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι εναντίον αυτής της μορφής βοήθειας. Πρέπει όμως οι βοήθειες αυτές να μην συνοδεύονται από κάποιες μορφές κινδύνου. Πάρα πολύ συχνά αυτοί που ωφελούνται από τις βοήθειες αυτές είναι όπως είναι φυσικό τρίτες χώρες. Τώρα εδώ πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Χώρες οι οποίες δεν έχουν ένα απόλυτα αναπτυγμένο δημοκρατικό σύστημα ελέγχου. Και είναι επίσης χώρες οι οποίες εν πολλής απειλούνται από την διαφθορά και ελέγχονται για περιπτώσεις διαφοράς πάρα πολύ συχνά. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τους κινδύνους αυτούς και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τους μηχανισμούς οι οποίοι να δώσουν e, Λοιπόν, ε, έχει επίσης ε, δοθεί και μία σύσταση προς, ε, την, ε, προς το ελεγκτικό συνέδριο έτσι ώστε να υπάρξουν περισσότερες στο μέλλον ειδικέ εκθέσεις σχετικά με θέματα που άπτονται της ε, άμεσης στήριξης από τον προϋπολογισμό. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία φάση επεξεργασίας 11 ειδικών εκθέσεων Δύο από αυτές τις τέσσερις σε μία πρώτη φάση εκθέσεις αφορούν την άμεση βοήθεια που δίδεται από τον προϋπολογισμό προς χώρες της Ασίας όπως επίσης και προς τον Ανατολικό Κάφκασο. Ελπίζω οι δύο αυτές εκθέσεις να είναι χρήσιμες έτσι ώστε να απλουστευτεί όσο περισσότερο γίνεται το μέσο αυτό το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Συγγνώμη λέει ο Πρόεδρος, ο εκπρόσωπος συνεδρίου, ξέχασα κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Είναι η τελευταία παρουσία μου εδώ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, να ευχαριστήσω όλους ε, τους ε, ευρωβουλευτές που ασχολήθηκαν με την υπόθεση αυτή. Χαίρομαι για το ενδιαφέρον αυτό. Οι συναντήσεις τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα ήταν ελπίζω χρήσιμες και για σας αλλά κυρίως για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για την προετοιμασία ε, των, της λειτουργίας ε, του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Σάικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επανέλθω σε ορισμένα σημεία τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί. Πάνω. Είμαστε στο 10ο ΦΕΤ και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ε, έξι ή επτά προτάσεις ε, ε, να εγγραφεί στο δημοσιονομικό, το κανονικό πλαίσιο, το ΦΕΤ, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει γίνει δεκτό. Θα το ξανακάνουμε φέτος, αλλά είναι σαφές να βρεθούν τα χρήματα και να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να μην υπάρχουν προβλήματα, για να μειωθούν μάλλον τα προβλήματα. Πάντα το υποστηρίζαμε και συμφωνούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς αυτό. Σχετικά τώρα με τις λεγόμενες εύθραυστες χώρες. Υπάρχουν πάρα πολλά συστήματα τα οποία ε, θα έλεγα στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί φυσικά και προσπαθούμε να βοηθήσουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση στην IT και κάποιες άλλες χώρες στα πλαίσια του ΕΚΟ το οποίο έχει κάποια συστήματα πιο ευέλικτα από τα δικά μας σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου. Υπάρχουν επίσης και άλλα συστήματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις καταστάσεις ε, οι οποίες ε, δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των κρίσεων ή μετά από αυτές. Σεβόμεθα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σειρά από κανόνες που μας επιτρέπουν να λειτουργήσουμε πιο ευέλικτα σχετικά με ό,τι έχει σχέση με τις ε, δημόσιες προμήθειες κτλ. Πολλές φορές μας κατηγορούν ότι οι διαδικασίες μας είναι πολύ ε, αργές. Δεν είναι εύκολο βέβαια να δημιουργηθούν σωστές διαδικασίες σε χώρες όπου δεν υπάρχει ο ανταγωνισμός, σαν παράδειγμα. Αλλά προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις. Επίσης ασχολούμεθα με τις κατευθυντήριες γραμμές για δημοσιονομική στήριξη προς τις εύθραστες λεγόμενες χώρες. έχει ακουστεί πάρα πολύ κριτική από πλευράς ε, του ελεγκτικού συνεδρίου για τις άμεσες αυτές βοήθειες. Να θυμίσω ότι η κριτική ε, του συνεδρίου είναι τυπική θα έλεγα, δεν είναι επί της ουσίας, δεν είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το συνέδριο πολλές φορές μας κατηγορεί ότι δεν τεκμηριώνουμε πάρα πολλές φορές τις δαπάνες αυτές. Νομίζω ότι η τεκμηρίωση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως είναι ιδιαίτερα αναλυτική. Υπάρχει πάντα μια ουσιαστική ανάλυση για τον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται ορισμένες δημοσιονομικές βοήθειες σε χώρες και υπάρχει η απαραίτητη τεκμηρίωση εν πάση περιπτώσει. Προφανώς και εργαζόμεθα ε, δραστηριοποιούμεθα σε χώρες οι οποίες παρουσιάζουν κινδύνους. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα προβλήματα δεν θα υπήρχε η βοήθεια για την ανάπτυξη. Και τα δύο πηγαίνουν μαζί. Πρέπει λοιπόν να προσπαθούμε να αξιολογούμε τους κινδύνους σε σχέση με αυτό το οποίο πρέπει να πετύχουμε. Και εδώ σε επίπεδο δημοσιονομικής βοήθειας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι δεν εργαζόμεθα μόνοι μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκεί όπου χορηγείται βοήθεια δημοσιονομική, συνεργάζεται με άλλους δωρητές, με χώρες μέλη επίσης, οι οποίες κάνουν το ίδιο. Συνεργαζόμαστε επίσης και ε, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα. Υπάρχει μια πραγματική συνεργασία και ε, θα έλεγα η συνεργασία αυτή είναι και σε επίπεδο λεπτομεριών. Σχετικά με τους ε, διεθνείς οργανισμούς έχουν υπάρξει ορισμένες αδυναμίες στα πλαίσια της συμφωνίας πλαίσιο με τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπεται να μας επιτρέπουν να ελέγχουμε ορισμένα εσωτερικά τους έγγραφα. Ε, σχετικά με την προσπάθεια την οποία εμείς κάνουμε ε, δεν μας δόθηκαν τα έγγραφα αυτά εγκαίρως και υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει επίσης μια αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής. Υπήρξε μια αποστολή της Επιτροπής σας η οποία επέτρεψε ε, να ε, λυθούν κάποια από τα προβλήματα και σχετικά ε, με την προσπάθεια που σε αυτή τη φάση κάνει το ελεγκτικό συνέδριο οι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΙΕ έδωσαν τα στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι υποστηρίζουμε το ελεγκτικό συνέδριο έτσι ώστε να είναι ικανό να λειτουργήσει σωστά σχετικά με τον έλεγχο των διεθνών οργανισμών. Όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα έχουμε, πάρει, ε, έχουμε παίξει το ρόλο μας και έχουμε βοηθήσει τη διαδικασία. Όταν το ελεγκτικό συνέδριο δεν έχει στη διάθεσή του τα παραστατικά που απαιτούνται, αυτό μας λυπεί Συνεργαζόμαστε με το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών και με το γραφείο τους εδώ στις Βρυξέλλες για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία είναι γενικά απλά και ελπίζω να επιλύονται στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχουμε σταδιακά βελτιώσει τη συνεργασία μας με τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πρέπει να κατανοούν και αυτοί το τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε και να κάνουν ό,τι χρειάζεται έτσι ώστε να γίνουν σεβαστές οι συμφωνίες που έχουμε συνάψει μαζί τους. Ολμέγερ έχει ζητήσει εκ νέου το λόγο. Απευθύνω εκ νέου παράκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην ωρεοποιήσει το θέμα των δημοσιονομικών ενισχύσεων που δίνει σε διάφορες χώρες. Μετά από τις συζητήσεις που έκανα με το ελεγκτικό συνέδριο και ακριβή ανάγνωση της έκθεσης, δεν μπορεί να πει κανείς ότι η έκθεση δεν αναφέρει παρά μόνο μικρά περιθωριακά σφάλματα τύπου φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές δυσχέρειες οι οποίες παρακολουθούνται από ετών που απασχολούν από ετών το ελεγκτικό συνέδριο εγώ βέβαια αυτά τα πράγματα τα βλέπω πρώτη φορά έχει υπάρξει απόκληση απόψεων και μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής με ανισχύει λοιπόν λίγο που η Επιτροπή μιλεί μόνο για δευτερεύοντα μικρά αμεληταία σφάλματα φαίνεται να μην συμβαδίζει αυτό απόλυτα με την πραγματικότητα. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να πάψετε να ωρεοποιείτε τα πράγματα στα θέματα των δημοσιονομικών ενισχύσεων. Οι δημοσιονομικές ενισχύσεις έχουν τα προβλήματά τους. Οι χώρες που τις δέχονται έχουν προβλήματα. Και επειδή έχω ασχοληθεί με τις χώρες αυτές γνωρίζω ποια είναι τα προβλήματα. Μην τα διατυπώνεται λοιπόν τόσο ελαφρά την καρδία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ για να ολοκληρώσει. Ε, Ξέρω τον κύριο Ολμάγερ, τα έχουμε ξαναπεί και καταλαβαίνω που το πάει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά η γνωμοδότηση του Ελληνικού Συνεδρίου απετέλεσε ε, κάτι πάρα πολύ θετικό μια που ε, μας λέει για τα πιο σημαντικά ότι, είναι όλα αξιόπιστα τα στοιχεία ε, με, με τις μικρές υποσημειώσεις επομένως ότι πρόκειτο παρά κάποιες λεπτομέρειες ε, πρόκειται για άρτιο οικονομικό έλεγχο μας ε, είχαν ανησυχήσει τα σκάνδαλα αλλά κατέβαλε προσπάθεια η Κομισιόν και έκανε έναν ε, κοσμητικό διάλογο με το ελληνικό συνέδριο κάτι το οποίο έλειπε το λέγαμε με τους συναδέλφους ότι θα πρέπει και με τη δική μου έκθεση επίσης να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι, ό,τι, ό,τι, ό,τι, ό,τι χρειάζεται και να τους ανταποδώσουμε επομένως με τη δική μας συμβολή το πόσο μας βοήθησαν. Βεβαίως και πάντα έχει σημασία το τι λέει το Ελληνικό Συνέδριο αλλά ιδίω αυτή τη φορά πέραν των επικρίσεων το κείμενο ήταν πάρα πολύ υποδομητικό. Ήταν και διδακτικό όπως και ο διάλογος με την Κομισιόν. Τετραγωνίσαμε τον κύκλο. Η ανεπτυξιακή βοήθεια είναι κάτι το επίγον, κάτι το αποτελεσματικό. Σε κάποιες ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες. και να λάβουμε πες υπόψη ότι ο δημοσιονομικός ένωσης δεν είναι πάντοτε εύκολος σε τέτοιες περιπτώσεις. Και τελικά μαζί με τον έρασμο η ανεψυχική βοήθεια είναι ό,τι προβάλλει καλύτερα την Ένωση στον κόσμο. Άρα τώρα μπορούμε να έχουμε διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στον έλεγχο του προπολογισμού και των λογαριασμών. Περιμένω και εγώ λοιπόν τις τροπολογίες των συναδέλφων. Θα συνεχίσουμε τη συνεννόηση, το διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεργαστούμε και με την νέα υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής. Οπότε να μπορέσουμε να δώσουμε νέα όθηση στα πράγματα με αφετηρία τη καινούργια υπηρεσία, καινούργια δομή. Ευχαριστούμε. Πέρα σα.